Bonjour et bienvenue. Χαίρετε και καλώ ήρθατε. Συνεχίζουμε τη χθεσινή συνεδρίαση. Ημερήσια διάταξη, σημείο 5. Απαλλαγή των λοιπόν θεσμικών οργάνων και καλώς ορίζω θερμά όλους τους γενικούς διευθυντάς και εκπροσώπους των λοιπόν οργάνων. Ο κύριο Ρούσο εξακολουθεί να απουσίας λόγω ασθενείας από το ηλεκτρικό συνέδριο θέλω να ζητήσω το εξή δεδομένου ότι τα υπόλοιπα μέλη δεν έχουν πάει για κυνήγι θα έπρεπε να αντικαθίσταται ένας ασθενής από κάποιο συνάδελφό του για χτες να το καταλάβω, για σήμερα δεν το καταλαβαίνω όμως και τελευταία εξαίρεση που δέχομαι γιατί απαιτώ να βρίσκονται εδώ οι παρόντες τα μέλη, παρόντα τα μέλη. Δέχομαι βεβαίως κανένα πρόβλημα να είναι το προσωπικό εδώ και οι συνεργάτες, αλλά δεν αντικαθίσταται ένα μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου από προσωπικό. Θέλω να μπορώ, να μπορούμε να διατυπώνουμε τις ερωτήσεις μας προς το ελεγκτικό συνέδριο για το ρόλο τους προς τα μέλη του. Δεδομένου ότι τώρα και σήμερα έχουμε μάλιστα την απαλλαγή του ελεκτικού Συνδρίου του ίδιου. Θα παρακαλώ τον κύριο Αλμπρίου να λάβει το λόγο. Τμήμα 5. Και σας διαβεβαιώ πώς πρόκειται και την τελευταία φορά που τον έχουμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. είμαι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Ευχαριστούμε που μας δίνεται το λόγο για να παρουσιάσουμε την ετήσια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου εκ μέρους του κυρίου Πιέτρο Ρούσου, για το 2017. Ο κύριος Ρούσο δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας. Το κεφάλαιο αυτό έχει να κάνει με την αξιολόγηση των δαπανών για όλα τα σώματα. Σε αυτό αναφέρεται 9,7 εκατομμύρια ευρώ ε, από το πολιτές νοσονομικό πλαίσιο και για το ελεκτικό συνέδριο έχουμε θετική αξιολόγηση χωρίς σημαντικό ποσοστό σφάλματος ε, βλέπουμε ένα 0,5% περίπου ποσοστό σφάλματος ε, για την ε, φετινή αξιολόγηση 55 ήταν οι συναλλαγές εκ των οποίων 12 που αφορούσαν το Συμβούλιο και 3 για το Συμβούλιο 3 για το Δικαστήριο Επιτροπή των Περιφερειών 2, ε, Ombudsman ένας Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ε, πάλι μία. Ε, συναλλαγή όπου συμπεριλαμβάνεται μία σχετική με σφάλμα ποσοτικά μετρήσιμο γιατί δεν είχε διατυπωθεί σωστά η κατάσταση για τις προηγούμενες μας συστάσεις. Η εφαρμογή γενική σύσταση για την διαχείριση μισθών και οικογενειακών επιδομάτων που είχαμε συμπεριλάβει στην ε, έκθεση του 2014 βλέπουμε να τηρείται πλήστον σε σχέση με τη σύσταση προς την ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ως προς την ε, διεξαγωγή δημοσίων προμηθειών. Θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση και σε περαιτέρω εξετάσεις, ε, και ελέγχους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας κυρίες και κύριοι. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ελέγχτε το δικαστήριο λοιπόν ο κύριος Βαλέιο Μπλάκο, Ζωμίσιο Λεχασέ, Βελέν Γουαρταρίκο. Η Γενική ο Γενικός Γραμματέας δεν είναι σε θέση να έρθει. Παρακαλώ, εσείς που ήσασταν και ασθενείς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας ε, προσκαλέσατε σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων ε, στην Επιτροπή. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Εξκομπάρ που δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα λόγω ακροαματικής διαδικασίας ε, ή στο πλαίσιο της επιταχυμένης ε, διαδικασίας που το άρθρο 50 ε, μια έκθεση για το Brexit. Έχουμε όμως τον κύριο Ρασέ, τον επιτετραμένο που είναι εδώ, να μας παρουσιάσει τα σχετικά. Το 2017 ήταν έτος στο οποίο το δικαστήριο ολοκλήρωσε τη δεύτερη φάση της ε, μεταρρύθμισης με τους δύο τελευταίους δικαστές που έπρεπε να οριστούν με ένα έτος καθυστέρηση συνολικά ως προς το χρονοδιάγραμμα και μένει ακόμα ένας δικαστής για να ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη φάση μεταρρύθμισης. Το 17 είχαμε δραστηριότητα 1668 υποθέσεις ε, και περί τις 1600 υποθέσεις φάκε, δηλαδή που έκλεισαν το δικαστήριο κατάφερε να μειώσει κατά 2,4 μήνες ε, την, τον μέσο όρο κάθε υπόθεσης σε περί τις 16 μήνες που είναι μια σημαντική μείωση σχετικά, μάλλον αναφορικά προς το έτος 2013. Το έτος είχε πολύ σημαντικές υποθέσεις ε, αρκετά ευαίσθητες. Εξεδόθησαν ε, αποφάσεις ε, στα πλαίσια του ασύλου της μεταναστευτικής κρίσης του 2015, και του κανονισμού για την κατανομή μεταξύ των κρατών μελών ε, των ετούντων άσυλο και της απόφασης Συμβουλίου 2015 σχετικά με τις ε, προσωρινές διευθετήσεις για, την, ε, για τον επαναπατρισμό. Επίσης εξετάσαμε την νομοποίηση των μαχητών της ISIS που έχουν επιστρέψει στις χώρες τους Κάποιο ενημέρωσε τον ομιλητή ότι μια είπε γρήγορα. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο ομιλητή. Λοιπόν, τώρα, σχετικά με τα δεδομένα των ε, επιβατών αερομεταφορέων στα πλαίσια της συμφωνίας ε, με τον Καναδά και ω προς την προστασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης είχαμε απόφαση σχετικά με τις υπηρεσίες της Uber, τις μεταφορικές υπηρεσίες. Εξετάσαμε επίσης την απόφαση της Επιτροπής ε, για πρόστιμο ενός δισεκατομμυρίου ε, σχετικά με μονοπωλιακές θέσεις ε, επιχειρήσεων. Επίσης, στα πλαίσια της κρίσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ή την διατήρηση της Χαμάς μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων, το καταλόγου δηλαδή. Αναπτύξαμε την ομολογία ή στην επιτήρηση των ε, τραπεζικών οργανισμών στην Ευρώπη μέσω δύο αποφάσεων διευκρινίσαμε την εποπτεία αυτή σχετικά με τις συγκεντρώσεις ε, τραπεζικών οργανισμών σε συγκεκριμένους ε, τομείς. Με την ομολογία αυτή λοιπόν εξετάσαμε πολύ ευαίσθητους τομείς, πολύ ευαίσθητα πεδία και βεβαίως πάντα εντός ε, του πλαισίου επιταχυμένης διαδικασίας ε, και λοιπόν υποχρεώσεων και πιο συγκεκριμένα την αδυναμία διαχείρισης των μεγάλων του αυξημένου όγκου εισρώων και την υποχρέωση εξέτασης ε, υποβολών φακέλων σε οποιοδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έτος 2017 επίσης σημειώθηκε από την δημιουργία του δικαστικού δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολυγλωσσικού δικτύου, που ενώνει τις δικαστικές αρχές των κρατών μελών και που, των οποίων το δικαστήριο αναλαμβάνει τον συντονισμό. Το δίκτυο αυτό είναι επιχειρησιακά έτοιμο από, το, από την αρχή του 2018, 18 επιτρέπει μια ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό των ομολογίων των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, δώσαμε παρακολούθηση στη σύσταση του ελεκτικού συνεδρίου για τον έλεγχο των δικαστικών υποθέσεων στα πλαίσια ενός νέου συστήματος διαχείρισης, το οποίο θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητά μας στη διαχείριση αυτή όπως είχε προβλέψει και το ψήφισμα για την απαλλαγή του 16. Επίσης, όπως προέβλεπε το ελεγκτικό συνέδριο, συνδέσαμε την ε, διάρκεια της εξέτασης της κάθε υπόθεσης με την περιπλοκότητα του θέματος καταφέραμε να διατηρήσουμε, να συγχωρείτε, την παραγωγικότητά μας με τη βελτίωση κάποιων μεθοδολογιών της εισρωής ε, σχετικό, ε, συγκεκριμένων εγγράφων και του e που το 2017 χρησιμοποιείται πλέον, χρησιμοποιήθηκε πλέον από όλα τα κράτη-μέλη και που είναι υποχρεωτικό από το Δεκέμβριο, αν ακούσαμε 18. περιορίσαμε το άχθος το μεταφραστικό στο 1,1 εκατομμύριο σελίδες ενώ το 2017 ήταν κατά 400.000 σελίδες ανώτερο το άκθος αυτό. Επίσης, διατηρήσαμε την ε, οριζόντια τη δυνατότητα των επιμέρους ε, ε, γραφείων μέσα στα πλαίσια της, ε, των αλλαγών στο προσωπικό που είχαμε. Επίσης, καταφέραμε να ε, αυξήσουμε τον αριθμό των φακέλων που κλείνονται κατά μέσο όρο σε 30% παρά τις περικοπές προσωπικού. ήμασταν στο 98,7% της απασχόλησης ε, σε ανώτατα επίπεδα, δηλαδή συνολικής απασχόλησης για το προσωπικό, δηλαδή χρησιμοποιούμε ε, στο 100% τα μέσα και το προσωπικό που έχουμε στη διάθεσή μας. Το 17 είχαμε, προχωρήσαμε και στην ε, αντικατάσταση 17 θέσεων και παγώσαμε επίσης τις δαπάνες ε, οι οποίες ε, αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% του συνολικού προϋπολογισμού των τρεχόντων εξόδων μας. Ε, τα στοιχεία δείχνουν τις προσπάθειες που κατέβαλε το δικαστήριο το 2017 και σε μία περίοδο από το 10 στο 17 επί τη βάση των συστάσεων του ελεκτικού συνεδρίου Επίσης ε, αυξήσαμε τις, ε, την ποσόστοση, το μέρισμα των γυναικών ε, στις θέσεις των υπαλλήλων και είχαμε και μια ομάδα εργασίας του 17 η οποία εργάζεται ώστε να άρει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν ίσως κάποιες φορέ οι γυναίκες προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε υπαλληλικέ ε, θέσεις συγκεκριμένου επίπεδου. Και για να προωθήσουμε την υποψηφιότητα τις γυναικείες υποψηφιότητες σε τέτοια επίπεδα. Νομίζω ότι συνολικά έχουμε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα ε, ε, σε άλλα πεδία όπως ε, το, τη μείωση του ίχνους του άνθρακα συνολικά για το όργανο. Επίσης αναπτύξαμε μια πολιτική εξωτερικής επικοινωνίας προκειμένου να προσεγγίσουμε τους πολίτες, ιδιαίτερα την νεολαία, με νέες μεθόδους επικοινωνίας ιδιαίτερα λογαριασμό Twitter και αρκετές, ε, αρκετά βίντεο στο YouTube τα οποία εξηγούν την όλη δραστηριότητα του οργάνου. Σας βεβαιώνουμε, Πρόεδρε, ότι θα εξακολουθήσουμε την προσπάθειά μας ε, βελτιστοποίησης αποτελεσματικότητας ώστε να αντιμετωπίζουμε το συνεχές άκθος ε, εργασίας που έχουμε Επίσης ε, για τη διόρθωση κάποιων υλικών λαθών για το ερώτημα 33 σχετικά με τις ασθένειες και τις απουσίες ε, τα έχουμε υποβάλει. Είμαστε διάθεσή για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. Καλώς ευχαριστώ και πάλι το, το δικαστήριο και για τη γραπτή απάντηση σε όλα μας τα ερωτήματα. Ελεκτικό συνέδριο τώρα λέει η Πρόεδρος. Όχι, η κυρία εισηγήτρια έχει τώρα η κυρία Χλαβάκοβα. κυρία Αγιάλα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν είχα καταλάβει ότι θα είχαμε διάλογο στο τέλος και θα ακούγαμε πρώτα όλους τους διευθυντές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο συνάδελφος ε, δεν μπορούσε να είναι εδώ, είναι ασθενή. Στο συγγνώμη εκ μέρους του μου ζήτησα να τον αντικαταστήσω για σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω το δικαστήριο για τις πληροφορίες που μας έδωσε σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των υποθέσεων υπάρχει το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων πλέον και το e-Courier και αυτά τα εργαλεία σίγουρα βελτιώνουν τη διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων, ωστόσο θα ήθελα να μου πείτε γιατί, ε, μάλλον τι αντίκτυπο έχει καθυστέρηση της ε, απόφασης στο πλαίσιο της ε, μεταρρύθμισης του δικαστήριου τριών δικαστών Δηλαδή δεν ορίστηκαν τρεις δικασίες, καθυστέρησε ορισμός των δικαστών. Τι ε, πτώση είχε σε ό,τι αφορά ε, τις υποθέσεις. Και θα μας ενδιαφέρει και κάτι ακόμη. Η απουσία δικαστών ε, στο πλαίσιο των λεγόμενων δικαστικών διακοπών, πώς επηρεάζει. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που είναι σε επιφυλακή ε, και αυτό πώς επηρεάζει τη διαχείριση των υποθέσεων. Ο κύριος Κοντ θεωρεί ότι η απάντηση στην ερώτηση 40 δεν δίνει το νούμερο που χρειαζόμασταν. Σε ό,τι αφορά το νέο κώδικα συμπεριφοράς για τα μέλη και η εκπόνηση κανόνων για το προσωπικό σε σχέση με τις περιστρεφόμενες πόρτες, μετάβαση δηλαδή από δημόσιο ε, οργανισμό σε ιδιωτικό τομέα. Θα ήταν καλοδεχούμενο να έχουμε και από αυτόν. Και τέλος μια ερώτηση για το πώς αναπτύσσεται μεταξύ των θεσμών αλλά ιδίω σε ό,τι αφορά το δικαστήριο, αν έχει πληροφορίες δηλαδή σχετικές, σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας στο Λουξεμβούργο. Να είναι πιο ελκυστικό το Λουξεμβούργο. Διότι το επίπεδο το βιωτικό εκεί, η μισθή καταβάλλονται σε σχέση με τις Βρυξέλλες φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο ελκυστική. Γνωρίζουμε πως υπάρχει διάλογο μεταξύ των θεσμικών οργάνων που έχουν την έδρα του στο Λουξεμβούργο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο συμπέρασμα προς το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η ελκυστικότητα των ε, θέσεων εργασίας στο Λουξεμβούργο και να αποφευθεί αυτή η μενεκτική θέση στην οποία βρίσκονται σε σχέση με το βιωτικό επίπεδο στις Βρυξέλλες. Και τέλος, Διεξοδικά μας μίλησε ο εκπρόσωπος ε, του δικαστήριου για το προσωπικό, για τις προσπάθειες που χρειάστηκε να γίνουν για τις περικοπές δηλαδή λόγω της συμφωνίας λιτότητας ε, στο θέμα των μισθών και του προσωπικού. Όμως οι 215 υπότροφοι που δεν αμείβονται ε, κάπως δεν μας φαίνεται και τόσο αποδεκτό στους αριθμός για το 2019. 550.000 ευρώ έχετε βάλει για τις υποτροφίες. Και ο κύριος Κοντ ρωτά, με αυτό τον αριθμό, με αυτό το ποσό, μήπως θα μπορούσε να εξασφαλιστεί και εξωπρεπής αμοιβή των υποτρόφων. Ευχαριστώ. Εσείς έχετε το λόγο, αλλά παρακαλώ να είστε σύντομος, διότι έχουμε το γύρο με τον σκιωδών εισηγητών και έχουμε και άλλους μετά που έπονται. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο της καθυστέρησης με τον ορισμό τριών δικαστών, ε, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των υποθέσεων, είναι απλά, απλή σχετικά η απάντηση. Αν είχαν οριστεί εγκαίρως οι εν λόγω δικαστές, η δραστηριότητα των του τμήματων θα ήταν πιο εντατική παρά βεβαίω την ανάγκη αυτό να σχετιστεί με την αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων γιατί είχαμε 24 ε, νέες αφήξεις μεταξύ της μερικής ανανέωσης και της μεταρρύθμισης της δικαστικής ε, αρχιτεκτονικής. Χρειάστηκε λοιπόν σημαντική δουλειά αναδιάρθρωση των τμήματων, ε, των δραστηριοτήτων και μετά το σχηματισμό τριών γραφείων με καθυστέρηση σίγουρα επηρεάστηκε ο ρυθμός εργασίας του δικαστηρίου όμως παρόλα αυτά οι διαδικασίες μειώθηκαν, η διάρκειά τους δηλαδή όπως προείπα, και το, τα διευρωμένα τμήματα που εδώ και χρόνια δεν λειτουργούσαν ξανά άρχισαν να λειτουργούν. Σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο από την απουσία δικαστών στη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, πολλές φορές το έχουμε εξηγήσει στην Επιτροπή σας, σε αυτές οι δικαστικές διακοπές και βάζω μέσα για τις λευκές εβδομάδες, όπως τις λέμε, δηλαδή που δεν έχουν ακροματικές διαδικασίες, Ουσιαστικά δεν είναι ε, διακοπές, δεν είναι άδεια περίοδος ε, αργίας. Απλά θέλουμε να εξορθολογήσουμε τη δικαστική δραστηριότητα. Γι' αυτό οι ακροματικές διαδικασίες ε, μόνο αν υπάρχει κατεπήγον οργανώνονται αυτές τις εβδομάδες σε συντονισμό με τις πρακτικές που υπάρχουν και στις εθνικές νομιστάξεις. Στόχος είναι η δικαστική λειτουργή και οι άλλοι πάλι να μπορούν όλοι μαζί ε, να αποφεληθούν ε, της διακοπής ε, επακροτηρίου διαδικασιών γιατί αλλιώς θα ήταν πολύ πιο πολύπλοκη η διαχείριση αν κάποιος δικαστής έλειπε κάποια συγκεκριμένη εβδομάδα να παρέλυαν οι εργασίες του συγκεκριμένου τμήματος το οποίο προείδρευε. Γι' αυτό τα έχουμε συγκεντρώσει. Δεν θα πει αυτό βέβαια ότι δεν εργάζονται δικαστέ ή ότι δικήν την περίοδο δεν βρίσκονται στο Λουξεμβούργο, διότι μονίμω εργάζονται οι δικαστέ, ακόμη περισσότερο και από του λοιπού υπαλλήλου. Ε, είτε βρίσκονται σπίτι του, ε, είτε στην έδρα του, στο γραφείο του. Ε, μόνιμα εργάζονται. Δεν υπήρξε αντίκτυπος, δεν υπάρχει αντίκτυπος, γιατί σε αυτά τα χρονικά διαστήματα οι δικαστές αν είναι στη δουλειά τους, μπορούν να συγκεντρωθούν στο να προχωρήσουν τους φακέλους που τους έχουν ανατεθεί ως εισηγητές και δεν τους διακόπτει από το έργο τους η ανάγκη να παρίστανται σε κάποιες ε, μακροτήριο διαδικασίες. Ε, τώρα, υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο ε, σε ό,τι αφορά τους ε, υποτρόφους και τις εξωτερικές ε, δράσεις. Για τις αρχές του 18, συγγνώμη, του 19. Για τις θέσεις στο Λουξεμβούργο Ε, συγγνώμη, αυτό που εννοούσα πριν δεν ήταν για τους υποτρόφους αλλά για τις περιστρεφόμενες πόρτες που είπατε. Ε, για το κόστος ζωής, πράγματι η κατοικία ανακριβή, η υγειονομική περίθαλψη. Ε, ε, υπάρχει μια διαβούλευση μεταξύ των θεσμικών οργάνων που έχουν έδρα στο Λουξεμβούργο. Και μάλιστα εγκρίθηκε μια έκθεση από μια ομάδα προβληματισμού με 24 συστάσεις. Στόχος η βελτίωση ε, της ε, ζωής των επαλλήλων και λοιπόν μελών να είναι πιο ελκυστικές θέσεις εργασίας, να υπάρχει ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και για τους νέους αποφύτους πανεπιστημίων. Υπάρχουν ε, ιατρικές περτιμολογήσεις και διάφορα άλλα ζητήματα. Θέλουμε όμως να προωθήσουμε, να προβάλλουμε και τα πλεονεκτήματα της ζωής ε, και της εργασίας στο Λουξεμβούργο. Υπάρχουν ε, μέτρα και για τη στέγαση και για τα κοινωνικά, στο κοινωνικό επίπεδο. Και τώρα αυτή η ομάδα είναι μια ομάδα παρακολούθησης που σε συντονισμό με τις άλλες ε, ε, ομάδες ε, εργασίας θα προχωρήσει τις εργασίες της. Υπάρχουν και οι μη αμοιβόμενοι ασκούμενοι. 505.000 έχουμε ζητήσει για το 19 για να έχουμε και στα γραφεία των δικαστών αμοιβόμενε περίοδους άσκησης, Γιατί μέχρι στιγμή μόνο στις υπηρεσίε μπορούσε να γίνει αυτό. Θα βελτιωθεί, πιστεύουμε, λοιπόν, το σύστημα. Θα έχουμε αυτέ τι αμοιβόμενε περιόδους άσκησης, αλλά με βάση τον περιορισμένο προπολογισμό που έχουμε. Και το σύστημα αυτό θα αρχίσει να εφαρμόζεται, απλά περιμένουμε να εγκριθεί ο προπολογισμό για το 2019. Και η απόφαση που θα αναδιατυπώνει τον κανονισμό για τις ε, περίοδους άσκησης ε, θα εγκριθεί και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά ισκιώδης, ε, παρακαλώ. Κύριο Αλαφράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω το δικαστήριο. Πράγματι, είδαμε και διαπιστώσαμε ότι ο των υποθέσεων αυξήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου το 16 το 17 σε σχέση με το 16, δηλαδή 1656. Το 16 όμως είχαμε 1628 υποθέσεις και το 17 1594 είναι υποθέσεις που επιλύθηκαν. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. και σε ό,τι αφορά την επίλυση ε, είχαμε μια, ένα περιορισμό της ε, διάρκειας. Αλλά πάντα και το 16 και το 17 σημειώνουν αύξηση σχέση με το 15 που είχαμε το χαμηλότερο, στο 16,1 ώρες, ε, μήνες. Οι πληροφορίες είναι πλήρη σχετικά, αλλά τι γίνεται με το Twitter και το YouTube. Δεν έχουμε επαρκή στοιχεία. 6. Ερώτηση 6 για το Brexit. Δεν μας δίνεται κανένα νούμερο. Και σε σχέση με τον ερώτηση 22, υπάρχουν 63 Βρετανοί που εργάζονται σε όλες τις κατηγορίες για το δικαστήριο. Έχει κάποια συγκεκριμένη πρόβλεψη για αυτά τα άτομα, 63 Τάνος υπηκόους που εργάζονται το δικαστήριο. Και τελευταία ερώτηση. 41 ερώτηση. Συζητούμε κάποια δεδομένα για τον ορισμό ειδικού συμβούλου για το Brexit και λέει deadline, αριθμός ενδιαφερομένων, ε, δημοσιοποίηση της ε, ε, προκήρυξης κτλ. Αλλά δεν μας έχετε απαντήσει σε καμία από αυτέ τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Κολέγη Vorsitzende. Κύριος Κλίντς, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα καταρχάς να κάνω μια γενική διαπίστωση. Χαίρομαι που με μία μόνο εξαίρεση έχουμε παρόντες όλους τους γενικούς γραμματείς εδώ. Βεβαίως αυτό καθιστά ακόμη πιο επώδυνη την απουσία του Συμβουλίου που όπως και πέρσι έκρινε ότι δεν είναι σκόπιμο να είναι παρόν εδώ. Εν πάση περιπτώσει όμως, τελευταία πεθαίνει η ελπίδα. Μπορούμε να το δούμε την επόμενη χρονιά. Και θα ήθελα να εστιαστώ στις συνέπειες του Brexit, γιατί είπατε ότι έχετε έναν ειδικό σύμβουλο, ο οποίος θα σας βοηθήσει να διατυπώσετε, να συντάξετε τα ιδιαίτερα μέτρα. Βέβαια αυτό σημαίνει πολύ περισσότερη δουλειά για σας στο μέλλον. θα καθαστούν απαραίτητες κάποιες δύσκολες αποφάσεις λόγω της ε, αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα δεν ξέρουμε πώς θα ολοκληρωθεί, πώς θα πραγματοποιηθεί αυτό το Brexit. Θα είναι μια συμπεφωνημένη αποχώρηση, θα γίνει χωρίς συμφωνία, πάρα πολύ πιο δύσκολα. Καλό θα ήταν λέει, να δούμε κάποιες ε, λεπτομέρειες για να μπορούμε να αξιολογήσουμε και τις συνέπειες μπορεί να έχει σε όρους οικονομικούς και κυρίως στις αμοιβές, α, και στις αμοιβέ των ασκουμένων ήδη ε, έγινε αναφορά. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς είναι δυνατόν να υπάρχει χωρίς αμοιβή ασκούμενο στο ελεγκτικό συνέδριο. Θα ήταν δείγμα κακοδιαχείρισης κάτι τέτοιο και θα ήθελα να ε, βεβαιωθούμε ότι δεν πρόκειται να συνεχιστεί. Παρακαλώ κύριος Γιάννη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα περιοριστώ στα δύο λεπτά οι δυνατόν. Καταρχά, θα ήθελα να κάνω παρατήρηση προς ε, απευθυνόμενη στο Συμβούλιο για να τονίσω για άλλη μια φορά πώ συνεχίζονται τα προβλήματα ω προ την διαφάνεια των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και επίση ότι θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή μα έχει δυσκολίε ε, στη διαδικασία τη απαλλαγή διότι δεν υπάρχει ικανοποιητική συνεργασία με το Συμβούλιο. Για άλλη μια φορά λοιπόν θα τονίσω πως χρειάζεται συνεργασία και πνεύμα ε, ανοιχτό από πλευρά του Συμβουλίου. Τώρα, θα ήθελα να τοποθετηθώ σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την ε, καθίδρυση ενός προσωρινού δικαστή στο δικαστήριο, προβλήματα συγκρούσεως συμφερόντων, και γενικά θα ήθελα να ξέρω τι συνέβη, τι μέτρα εισήχθησαν σε επίπεδο δικαστηρίου για να απαφευθούν προβλήματα τέτοιου τύπου στο μέλλον, δηλαδή συγκρούς συμφερόντων, όπως αυτή που είδαμε στην περίπτωση του κυρίου Ταράγκας, για το ελεκτικό συνέδριο. Ο κύριος Πίνξταν, πρώην μέλος και από αυτά που μας λέει και η έκθεση της Όλαφ στην υπόθεση αυτή. Φαίνεται να υπάρχουν εδώ πέρα πάλι κάποια, ε, να υπάρχει απουσία συστημικών ελέγχων ε, σε επίπεδο ελεγκτικού συνεδρίου και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σκοπεύετε να κάνετε για να επαναφέρετε ελέγχους ικανοποιητικού ώστε να αποφευχθούν οι πρόεδρος. Μα κάναμε διαφοροποίηση σε σχέση με το ελεγκτικό συνέδριο. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε μόνο για το δικαστήριο. Κύριος Δε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λίγες ερωτήσεις έχω μόνο για το νέο κώδικα διοντολογίας ή τις ελλαγές. Νομίζω ότι πάμε στη σωστή κατεύθυνση, αλλά η ερώτηση μου είναι αντίστοιχη με του κυρίου Γιάργου. Πώς διενεργούνται οι έλεγχοι. Δηλώνουν τα οικονομικά και άλλα συμφέροντά τους στα κρατημέλη, αλλά αυτά ελέγχονται και επίσης προτού πάμε σε συγκεκριμένη εξέταση ελέγχουμε τη δήλωση του κάθε υποψηφίου και αρκούμαστε σε αυτό ή ψάχνουμε για κάποια άλλη ενημέρωση. Τώρα για, τις, ε, για τη μεταπίδηση στον ιδιωτικό τομέα και τις ε, περιστρεφόμενες πόρτες. όπως και για τις αποστολές έχουμε και εκεί κάποια ερωτηματικά σχετικά με τα ποσά που απαιτούνται αλλά πάντοτε το πρόβλημα ήταν ή ε, τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης στα οποία, τα οποία μάλλον παρακολουθούν οι δικαστές και ποια από αυτά είναι απαραίτητα για τα καθηκοντά τους και όχι, όχι. Αυτό ήταν, το ανέφερα ήδη. Αυτά είχα. Ευχαριστώ. Επειδή πρέπει να πάω και στη Γερμανία, και εγώ στον κατάλληλο των θα πάρω τώρα το λόγο. Τι γίνεται με αυτές ε, τις, ε, τα fuel cards και πώς ε, ε χρηματοδοτείται η οικογένεια, καλύπτεται ή όχι. Και το δεύτερο ερώτημα για το 56 το Μάη φέτος στην Πορτογαλία είχαμε το ε, συνέδριο αλλά πήγαν 12 διερμηνείς και σχεδόν 80 άλλοι δηλαδή 100 συμμετέχοντες ήταν όλοι όλοι είπατε ότι δεν δίνετε χορηγία αλλά αν έχετε 12 διερμηνείς μαζί οπωσδήποτε κάτι κάποια χρήματα δίνετε Σίγουρα ήταν ένα τεράστιο πάρτι, ε, υπαλλήλου με πολλούς εκεί παρόντες. Ποιος ε, και πώς τα πλήρωσε. Και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ε, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Θα αναγκαστώ να φύγω όμως ε, και θα με εκτεθεί ο κύριος Βόν και στο συγγνώμη των προτέρων παρακαλώ απαντήστε σε όλα αυτά. Je remercie. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, τα μέλη της Επιτροπής που έθεσαν μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με τη δραστηριότητά μας. Σχετικά με τον αριθμό των υποθέσεων που ελαφρά κατήλθε σχετικά με το 16, αυτό εξηγείται μέσω της ανάγκης αναδιοργάνωσης του δικαστηρίου μετά τις δύο πρώτες φάσεις της μεταρρύθμισης είχαμε την μαζική εισρωή νέων δικαστών χρειάστηκε να ενσωματωθούν αυτά τα νέα μέλη μετά την αναδιοργάνωση της δραστηριότητα ε, με διαφορετικές δηλαδή δομές οργανωτικές νομίζω ότι είναι κατανοητό χρειάζεται μια μεταβατική περίοδος προτού ας πούμε η μεταρρύθμιση αποδώσει πλήρως καρπούς της και η αναδιοργάνωση. Αλλά η βάση ρητώση η διάρκεια εξέταση των φακέλων ξεκάθαρα μειώθηκε όπως ήδη σας είπα και η σχέση, ο λόγος μεταξύ των φακέλων που κλείνουν και των συνολικών που υποβάλλονται είναι πολύ θετικός. Για το λογαριασμό Twitter έχουμε 53.000 followers, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Με πολύ υψηλό δείκτη δέσμευσης των followers αυτών, λέει ο ομιλητής. Επομένως υπάρχει σημαντικός αριθμός ανθρώπων που παρακολουθούν τις υποθέσεις αυτές Για τους ε, Βρετανούς συναδέλφους ε, τους 63 ε, στις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο είπαμε ότι ανακοινώσαμε ότι επί της αρχής θα χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν θα έχει επικότητα κράτους μέλους εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που θα είναι προς το συμφέρον του, της υπηρεσίας να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τους ανθρώπους αυτούς, οι υπόλοιποι θα πρέπει, τους ειδοποιήσαμε δηλαδή, ότι θα αποχωρήσουν. Ε, παρακολουθούμε διαρκώς το Brexit και τον ε, νομικό αντίκτυπό του υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που δεν εμφανίζονται στο ερωτηματολόγιο όπως τις διαδικασίες επιλογής. Δεν υποχρεωνόμαστε υπό το 123 να ακολουθούμε συγκεκριμένη διαδικασία ε, ανάρτησης, δηλαδή καινής θέσεως προ της διαδικασίας επιλογής, Είχαμε εξάλλου εξηγήσει ότι ο κύριος Μπράντλε που είναι ο ειδικός, ο σύμβουλος στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε προσληφθεί λόγω πολύ συγκεκριμένων δεξιοτήτων, ικανοτήτων που ήταν πολύ κοντά στα καθήκοντα που επρόκειτο να του ανατεθούν. εκτός φυσικά από την εμπειρία του που ήταν ε, πρώην δικαστής και επικεφαλής ε, της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για την προετοιμασία των ε, στάζ των... και μετά τον διαμεσολαβητή, την παρέμβαση του διαμεσολαβητή, εξετάσαμε προσεκτικά το θέμα και εδώ και αρκετά, αρκετούς μήνες έχουμε ένα σχέδιο απόφασης. Περιμένουμε απλώς τις απαραίτητες επιστώσεις από την αρχή προϋπολογισμού για τη σύγκριση συμφερόντων των μελών. Τα μέτρα που εισήχθησαν από τον κώδικα διοντολογίας, τα οποία ισχύουν ήδη, Δηλαδή ήδη εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά, δεν είναι ότι πρόκειται να αναλυφθούν ε, και θέτουν ένα πλαίσιο πολλαπλών υποχρεώσεων για τα μέλη. Σχετικά με το ποιος θα μπορούσε να υποβάλει ε, οποιαδήποτε ένσταση σχετικά με την αμεροληψία τους ή ακόμα και την αίσθηση, την εντύπωση της αμεροληψίας τους και έχουμε και πολύ συγκεκριμένε ε, λεπτομέρειες ε, σχετικά με τις επενδύσεις ε, ή αγορές τίτλων που μπορούν να έχουν προκειμένου να μπορούμε να έχουμε μια συγκριτική ανάλυση πριν τον ορισμό οποιασδήποτε υπόθεσης, οποιοδήποτε φακέλου για τα μέλη αυτά και προς αποφυγή οποιασδήποτε σύγκρουση ε, συμφέροντος. Υπάρχει πάντοτε και η δυνατότητα να μην συμμετάσχει συγκεκριμένο μέλος εθελοντικά εφόσον θεωρεί ότι υφίσταται τέτοια περίπτωση, τέτοια πιθανότητα. Για τις αποστολές ε, των μελών είχαμε εξηγήσει ότι αυτές επιτρέπουν στα μέλη να εκπροσωπούν το όργανο. Ε, κύριε Εσκοβάρη, πρέπει, πρέπει, έχετε μακρηγορήσει, πρέπει να συντομεύσετε. Ζητώ συγγνώμη. Ναι, ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε. Οι αποστολές είναι ουσιαστική ε, σημασία προκειμένου το δικαστήριο να είναι σε επαφή ε, με, τις, ε, με τα κράτη-μέλη από τα οποία προέρχονται τα μέλη του Έχουμε τα σχετικά μεγέθη κατανάλωσης, αλλά δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο επιβάρυνσης του προϋπολογισμού, λέει ο μιλτής. Και για το κεντρικό σύστημα διαχείρισης δεν, ναι, δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο πρόεδρε, εφόσον μου ζητάτε να συντομεύσω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ μεγάλη χαρά μου έδωσαν αυτά που είπατε για το προσωπικό σας για το Brexit. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ε, αν συνεχίσουμε όμως με τους ρυθμούς αυτούς θα μας πάει δύο η ώρα για να τελειώσουμε και θα σας παρακαλέσω να συντομεύετε. Μέχρι πέντε λεπτά παρακαλώ στην επόμενη ε, από, ε, από το ελεγκτικό συνέδριο. Έχουμε τον Ιανουάριο συνεδρίαση ε, με τον πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου για να συζητήσουμε το θέμα του Βέλγου που ήταν μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου και έτσι ξέροντας μεν ότι οι συνάδελφοι θα ήθελαν πολύ να κάνουν τις ερωτήσεις τους ε, παρακαλώ να, το, να τις ε, συγκρατήσουμε για την επόμενη ευκαιρία. Κύριε Γενική Γραμματέφετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ στα Ισπανικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους ευρωβουλευτές. Ε, το 2017 το Ελεκτικό Συνέδριο εκπλήρωσε την αποστολή του 93 δημοσιεύσεις, ε, δηλαδή μια ε, δημοσίευση κάθε τέσσερις θέσεις ετήσια έκθεση, 28 ειδικέ εκθέσεις, 55 αιτήσιες ειδικέ και διάφορες γνωμοδοτήσεις, αναλύσεις και ενημερωτικά έγγραφα. 50 εκατομμύρια 900 περίπου ημέρες, εργατοημέρες και πέρυσι 28 κράτη-μέλη ε, ελέγχθηκαν. Ε, επίσης επισκεφτήκαμε και 27 τρίτε χώρε και εστιάσαμε στους τομείς ε, ενδιαφέροντος για το Κοινοβούλιο που είναι η νεανική απασχόληση, συνδρομικές μεταφορέ, νέοι ουρανοί, διαχείριση πόσιμου ύδατο, νεαροί αγρότες ή μετανάστευση και hot spots συγκεκριμένα. Επίσης, δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στην οικονομική διακυβέρνηση και δημοσιεύσαμε για την ε, ελληνική κρίση ένα ε, εκείμενο, καθώς και για την ε, ενιαία, ενιαίο φορέα εξυγίανσης. Επίσης, ό,τι αφορά το δικαστήριο επίσης ε, δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή, όπως και στη σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος μας, ο κύριος Λέν, κατέθεσε το πρόγραμμα εργασίας και την ετήσια έκθεση ε, μαζί με τον κύριο Λάθαρο ε, και επίσης τα μέλη μας είχαν 60 παρουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχαν και πολλές διμερείς επαφές. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ καλή συνεργασία και έτσι μπορούμε νομίζω να βοηθήσουμε το Κοινοβούλιο προτρέχοντας, προκαταλαμβάνοντας τα αιτήματα και επίση δημοσιοποιούμε και πιο αποτελεσματικά έτσι τα αποτελέσματα των ελέγχων. Σε ό,τι αφορά του βασικού δείκτε αποτελεσμάτων, είναι θετική η κατάσταση, θετική εκτίμηση σε ό,τι αφορά την ποσότητα των εκθέσεων και αρκετά υψηλή αποδοχή των συστάσεων των εκθέσεων. Σε ό,τι αφορά την προβολή μα από τα μίντια, και εδώ έχουμε αύξηση, μεγαλύτερη προβολή το 2017 και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά στου πολίτε. Ήθελα να, να υπογραμμίσω ότι ε, το μέσος χρόνος ε, παραγωγής ε, των εκθέσεων 14,6 μήνες κατά μέσο όρο. Σίγουρα δεν είμαστε στους 13 μήνες ακόμη, όπως απαιτεί ο χρηματοοικονομικός κανονισμός, ο δημοσιονομικός κανονισμός και ξέρω ότι αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη δική σας επιτροπή το ηλεκτρικό συνέδριο συνέχισε να ανοίγει τις πόρτες του στον ακαδημαϊκό κόσμο με δύο στόχους, τη διαφοροποίηση και αύξηση της ε, ειδική γνώσης, των εξειδικευμένων γνώσεων, αλλά και προσέγγιση προς πολίτες και ιδίως στους πιο νέους ηλικία. Και ξεκίνησαν ε, έτσι διάφορες πρωτοβουλίες σε συνεργασία με διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια το 2017. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ο ρυθμός των ε, γυναικών που είναι στελέχη ε, principal manager ή directors ε, είναι γύρω στο 37%. Και βεβαίως ε, καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει έλλειψη ισορροπίας ακόμη, ιδίως ό,τι αφορά τους ελεγκτές. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουν τις προσπάθειες για βελτίωση. Πρόσφατα, το ελεγκτικό συνέδριο στο πλαίσιο ενός νέου σχεδίου για ισότητα ευκαιριών έθεσε ένα στόχο ποσόστοση του 40% για όλες τις θέσεις στελεχών που θέλουμε να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια. Το ελεγκτικό συνέδριο διαχειρίστηκε ε, με πολύ αυστηρό τρόπο τους ε, πόρους του, σε ό,τι αφορά τη μείωση του 5% του προσωπικού το ολοκληρώσαμε. Η δημοσιονομική εκτέλεση 98% έκταση του προπολογισμού, δηλαδή έκθεση εσωτερικών ελεγκτών και εξωτερικών ελεγκτών ήταν θετικέ. Βελτιώσαμε την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού και έχουμε και την περιβαλλοντική πιστοποίηση έμας. Άρα νομίζω ότι το 2017 το ελεκτικό εκπλήρωσε την αποστολή του να βοηθά το Κοινοβούλιο και ε, στην υποβολή των λογαριασμών και στην χρηστή διαχείριση. Επίσης, παγιώσαμε τις οργανωτικές μεταρρυθμίσεις που δρομολογήσαμε προσφάτως για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις νέες πολιτικές δαπανών, το νέο δημοσιονομικό ορίζοντα και τα νέα μέσα διαχείρισης ελέγχου και τα δημοσιονομικά νέα μέσα. Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων και το παράρτημα που σας έχουμε διαβάσει και απαντήσει στο ερωτηματολόγιο νομίζω ότι σας δίνουν πιο αναλυτικές πληροφορίες αλλά φυσικά είμαι και στη διάθεσή σας εφόσον θέλετε να μου υποβάλλετε κάποιο ερώτημα. Ευχαριστώ. Μπράβο σας και ίσα που δεν αγγίξατε τα πέντε λεπτά. Άι, αλλά σέντερ. Βεβαίω. Ευχαριστώ πολύ και πάλι, ε, κύριε Πρόεδρε αντικαθιστώ τον κύριο Κόντου που για λόγους υγεία δεν μπορούσε να είναι εδώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα, επειδή μας ενδιαφέρει πολύ, να μου πείτε λίγο περισσότερα πράγματα για τις ε, ε, διαπραγματεύσεις ε, με την Όλαφ για μια νέα διοικητική συμφωνία και επίσης με τη νέα Σαγγελική Αρχή. Ποια συνεργασία έχετε. Πώς προχωρούν διαπραγματεύσεις συμφωνίες. Έχουμε και την ε, ακρόαση, δεν θα πούμε σε λεπτομέρειε, αλλά ξέρουμε ότι υπήρξε βελτίωση, υπάρχουν και κάποιοι έλεγχοι που προβλέπονται. Σε ό,τι αφορά τις αποστολές, απουσία, παρουσία των μελών. Αυτή η μελέτη, αυτή η αναθεώρηση πότε θα γίνει, εγκρίνεται ε, από την Ολομέλεια. Κάτι τέτοιο. Εμείς παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά το θέμα αυτό. Επίσης, είπατε κι εσείς, υπάρχει θέμα με την ισότητα ανδρών και γυναικών για το προσωπικό, σε τον ορισμό των ελεγκτών, που και εκεί υπάρχει πρόβλημα. σε αυτή τη διαδικασία απαλλαγή θα πρέπει να υπενθυμίσουμε για μία ακόμη φορά στα κρατημέλη την ανάγκη να υιοθετήσουν μία διαδικασία ώστε να υπάρχει ισορροπία, ενα άντρα μία γυναίκα. Ώστε να υπάρχει τουλάχιστον 50% ε, γυναικείες υποψηφιότητες, 50% ανδρικές υποψηφιότητες. Είπατε ότι έχετε τώρα αυτή την ποσόστοση 40%. Φαντάζομαι ότι θεωρείτε με αυτή την ποσόστοση ότι μπορείτε να έχετε κάποια θετικά αποτελέσματα. Για πείτε μου όμως ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας. Γιατί εγώ θα έλεγα ότι ο στόχος μας είναι το 50%. Τέλος. Έχουμε ένα εκατομμύριο ευρώ για εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη, πραγματογνωμοσύνη τέλο πάντων, σε σχέση με την εξήγηση των τραπεζών. Έχει κατακριθεί αυτό ποσό. Μήπως καλύτερα θα ήταν αυτές οι δαπάνες να πάνε για ε, τους εσωτερικούς εμπειρογνώμονες, διότι ήρθε για να μείνει το θέμα των τραπεζών δεν είναι κάτι που θα περάσει, δεν είναι κάτι προσωρινό. Τέλος. Σύγκρουση συμφερόντων. Έχουμε αντιληφθεί κυρίως λόγω της επιλογής ή παραμονής κάποιων ελεγκτών ε, και της ε, επικέντρωσή σε συγκεκριμένα θέματα είναι κάπως σαν να, επιλέγουν κάποια θέματα με βάση τα προηγούμενα ενδιαφέροντα ή συμφέροντά τους. Και έχω εγώ τουλάχιστον στο μυαλό μου δύο περιπτώσεις, αλλά αν το μελετήσω σε βάθος και ε, σκαλίσω λίγο πιο βαθιά θα βρω κι άλλους φαντάζομαι. Πώς το ελεγκτικό συνέδριο σκέφτεται να αποφύγει τον να υπάρχει οποιαδήποτε ε, σκιά ε, υποψίας ε, για ενδεχόμενο σύγκρουση συμφερόντων. Γιατί έχετε να κάνετε με πάρα πολύ λεπτά θέματα και τώρα επεξεργαζόμαστε τον ε, ισολογισμό και τα αποτελέσματα. Αν δεν υπάρχει σαφής αμερόληπτη στάση και αντικειμενικότητα, όλα αυτά οδηγούν σε υποψίες και αμφιβολίες. Μήπως πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα των ελεγκτών για να μην ε, ε, κάθονται, πώς να το πω, στροκυλοκάθονται σε κάποια συγκεκριμένη αίθουσα και ε, εξειδικεύονται σε κάποια συγκεκριμένα θέματα. Και έτσι δεν είναι τόσο πια αμερόληπτοι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω ο γραμματέα. Γραμματέας. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να αρχίσω με την Όλαφ. Η συμφωνία προχωρά, είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να πω το εξή. Ακόμη και πριν αυτή τη νέα συμφωνία που διαπραγματευόμαστε και σύντομα θα την υπογράψουμε, η σχέση συνεργασίας με την Όλαφ ε, είχε συνεχίσει όπως και πριν. Πρόσφατα, για παράδειγμα, ε, διοργανώσαμε κοινέ ημερίδε επιμόρφωσης και ένα σεμινάριο ανταλλαγή πρακτικών ε, προβλέπεται για του χρόνου. Υπάρχουν κάποια κενά που θέλουμε να κλείσουμε σε ό,τι αφορά το ρόλο του Ευρωπαίου Αγγελέα. Ένα θέμα που θα το παρακολουθούμε πάρα πολύ σύνδεση και θα επηρεάσει την ε, Όλαφ ως προς το έργο της, αλλά και το ελεγκτικό συνέδριο Πώς δηλαδή θα επικοινωνεί για αυτές τις ε, υποθέσεις ενδεχόμενης ε, απάτης. Ε, Επομένω, όταν κλείσουν και αυτά τα κενά θα έχουμε τη συμφωνία και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και πιο αναλυτικά για τη σχέση που θα έχουμε και με τον Ευρωπαϊκό και με την Όλαφ στο μέλλον. Εν αναμονή βέβαια της, του καθορισμού της εντολής και του ρόλου του Ευρωπαίου Αγγελέας. Ό,τι αφορά το τέος με, μέλος του ελεκτικού. Δεν θέλω βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί αυτό θα γίνει στις 29 του μήνα, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Απλά θέλω να πω ότι ήδη από το 2016 το ελεγκτικό συνέδριο άρχισε να λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της ε, χρήσης ό,τι αφορά τους οδηγούς, τα αυτοκίνητα και τις αποστολές των μελών. Ιδίω το 2018 οι εγκρίσεις ε, ε, αποστολών για τα μέλη μέχρι το Φεβρουάριο του 2018 ήταν κάτι το οποίο το είχε αναλάβει ο πρόεδρος και το εκχώρησε στο Γενικό Γραμματέα. Όλες οι αποστολές πλέον εντάσσονται στο ίδιο σύστημα ελέγχου, όπως και οι υπόλοιπε αποστολές και υποβάλλονται τους ίδιους εσωτερικούς ελέγχους, εξάντε και εξπόστο. Επομένως, ε, ναι βέβαια και πριν ήταν ε, σε ισχύ έλεγχη, όμως τότε τις, ε, ε, το είχε αναλάβει αυτό το καθήκον ο πρόεδρος, τώρα θα το έχει ο Γενικός Γραμματέας και νομίζω ότι αυτό δίνει μια μεγαλύτερη ε, στεναρότητα στο σύστημα γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο ο έλεγχο, ε, πολύ περισσότερες οι περιπτώσει που πρέπει να ελεγχθούν και τώρα θα γίνεται αυτό με πιο μεγάλη αποτελεσματικότητα. Σε ό,τι αφορά την Όλαφ, ε, η έκθεση δεν αφορά συστημική, συστημικό πρόβλημα ε, στο ελεγκτικό, αλλά μια μεμονωμένη περίπτωση. Σε ό,τι αφορά την ισότητα ευκαιριών, σε ό,τι αφορά αυτή την ποσόστοση του 40%. Ποια ήταν η πρόθεση, ποια ήταν η ιδέα. Ήδη να πω βέβαια ότι αυτό το 40% ισχύει σε ορισμένα τμήματα. Είναι πραγματικότητα στη δίκη και στην μετάφραση. Και σε κάποια χαμηλότερα στελέχη, επίσης εκεί έχουν πάνω από 40% γυναίκες, το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε κυρίως στον τομέα των ελεγκτών. Ε, με βάση τον υπολογισμό που έχουμε, που είναι ένα κατά προσέγγιση βέβαια υπολογισμό, γιατί βασίζεται σε διάφορε υποθέσει και σενάρια, για το πότε θα συνταξιοδοτηθούν κάποιοι managers, κάποιοι διευθυντέ. Και σίγουρα έχουμε και πάντα το κριτήριο τη αξιοκρατία. Για το 2017-2019 θα μπορούσαμε να φτάσουμε, πιστεύουμε, στους 47% για την εξήγηση των τραπεζών. Το ελεγκτικό συνέδριο σε τρία μέτωπα κινούμαστε ταυτόχρονα. Το πρώτο, θέλουμε να αυξήσουμε την εσωτερική ε, εμπειρία και τις εσωτερικέ γνώσεις των υπαλλήλων. Γι' αυτό χρειάζεται ήδη να μάθουμε να λειτουργούμε ε, και να μάθουμε το αντικείμενο ουσιαστικά. Η εξήγηση τραπεζών, ευτυχώ γιατί δεν χρειάζεται να γίνουν πολλέ εξηγήσει, δεν είναι να ε, θέμα που, για το οποίο υπάρχουν πολλοί ειδικοί, πολλοί εμπειρογνώμονε. Οι δε περισσότεροι από αυτού που υπάρχουν προτιμούν, όπω είναι προφανέ να εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, άρα βρήκαμε δύσκολα εμπειρογνώμονε. Πάντω κάποιου του βρήκαμε, του έχουμε προσλάβει και οργανώνουμε και την εσωτερική επιμόρφωση. Αν χρειαστεί, ίσως ε, αναγκαστούμε να προσφύγουμε σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Αυτό θα βελτιώσει την κατάσταση, θα είναι καλύτερο ο έλεγχο που θα γίνει και αυτό θα μα δώσει και εμά τη δυνατότητα να αποκομίσουμε γνώσει ε, και εσωτερικά να μπορούμε πλέον να εργαζόμαστε καλύτερα. Σύγκρουση συμφερόντων. Δεν γνωρίζω τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω. Αλλά όπως γνωρίζετε, τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου πρέπει να κάνουν αυτή τη δήλωση ε, συμφερόντων, την οποία εξετάζει ο πρόεδρος ε, και βέβαια ε, πρέπει να τηρούν και κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς. Όποτε ένα μέλος θεώρησε ότι μπορεί να υπάρχει σε κάποια σύγκρουση συμφερόντων για την περίπτωση κάποιου συγκεκριμένου ελέγχου, απεσύρθη από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αν τώρα υπάρχει κάποιο πιο συγκεκριμένο ερώτημα, με τα χαράς να το απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γραμματεύ. Γενικέ Γραμματεύ. Σκιώδης με τον κύριο Σαλαφράνκα πρώτα. Ε, Είδαμε με ικανοποίηση το 2017 μέσο μέσος χρόνος από την έναρξη της, του ελέγχου μέχρι το τέλος ε, την εκπόσης έκθεση ήταν 14,6 μήνες και είναι το πιο σύντομο διάστημα για την περίοδο 2013-2017 σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις που δημοσιοποιήθηκαν 13 μήνες και λιγότερο ήταν ε, ε, μέχρι τη δημοσιοποίηση περίπου 17 μήνες λιγότεροι από το 2017 είναι θετική αυτή η τάση που δείχνει ότι τα μέσα τα μέτρα μάλλον για τους 12 μήνες που προβλέπει ο δημοσιονομικός κανονισμός ε, δίνουν καρπούς. Επίσης το 2017 το 65 των ειδικών εκθέσεων δημοσιοποιήθηκαν από το ελεγκτικό εντός προθεσμίας. Όμως ε, Σε ό,τι αφορά το ερωτηματολόγιο, θέλω να επιμείνω σε κάποιε ερωτήσει που νομίζω δεν έχουν απαντηθεί ικανοποιητικά. Η δεύτερη ερώτηση για τα κοινωνικά δίκτυα, όπω και για την περίπτωση του δικαστηρίου. Δεν έχουμε πληροφορίε για του ε, followers ή για, την, ε, για τα ποσοστά. Τι ποσοστά ήταν χρήσιμο για να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη απάντηση για το 2015. Τώρα ζητούμε πληροφορίε για τι ε, ε, επαμοιβή δραστηριότητες. Ούτε εδώ έχουμε κάποιον σε ό,τι αφορά την ερώτηση 33. Λέω ότι υπήρξε εσωτερική ανάθεση κάποιων δραστηριοτήτων για το μετριασμό των ε, επιπτώσεων της υποχρεωτικής ε, περικοπής του προσωπικού. Δεν μας λέτε τι συγκεκριμένα. Ε, είναι αόριστη απάντηση στην ερώτηση. Και τέλος, ερώτηση 37. Σε ό,τι αφορά τη μείωση των αποστολών γίνεται σύγκριση με το έτος αναφοράς 2014. Αλλά ε, το 17 είναι το έτος αναφοράς για την απαλλαγή. Δεν καταλαβαίνω γιατί χρησιμοποιείτε το 14 ως βάση. Ο κύριος Κλίντς είναι ο επόμενος. Ναι, στην έκθεσή σας μιλάτε για ένα πρόγραμμα ασφαλή χώρος εργασίας. Τι σημαίνει αυτό 1,7 εκατομμύρια, τι συνέπειες έχει, τι απόδοση έχει, είναι μόνο ένα ποσό κατά ή θα έχουμε επανάληψή του στον προσεχή προϋπολογισμό και επίσης το ελεγκτικό συνέδριο το ευρωπαϊκό, τι είδους συνεργασία ή σχέση έχει με τα εθνικά και λειτουργεί ως ε, κόμβος επικοινωνίας για την ανταλλαγή και διάθεση εισαλλήλους βέλτιστων πρακτικών. Υποστηρίζεται η πρόθεση του Κοινοβουλίου για την επιτάχυνση της διαδικασίας της απαλλαγής, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τηρήσουμε πιο απαιτητικά χρονοδιαγράμματα του χρόνου. Γιάβο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ε, θα προσπαθήσω κι εγώ να περιορίσω το χρόνο με, τις, με όλες τις ερωτήσεις που έχω για τα δύο όργανα σε δύο λεπτά μόλις. Ε, αν και υπάρχει αρκετό υλικό να συζητήσουμε με την ε, συγκεκριμένη υπόθεση, όπως είπατε και εσείς, στην κεκλεισμένα των φερών συνεδρίας που θα γίνει αργότερα. Κύριε Γκαρσία, εσείς είπατε ότι πρόκειται για μια μεμονωμένη υπόθεση και όχι συστημικό πρόβλημα. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ακριβώς ότι πρόκειται για μια μεμονωμένη περίπτωση και όχι συστημικό φαινόμενο. Ε, όταν υπήρχε αν υπάρχει συστημικός έλεγχος και αν αυτός ο συστημικός έλεγχος έχει δείξει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, τότε να πούμε ότι ήταν ε, μεμονωμένο το πρόβλημα της ε, παράτυπης συμπεριφοράς του συγκεκριμένου αυτού ε, μέλους, αλλά κατά τα άλλα θα παρακαλέσω να γίνονται τακτικά και συστημικά ή και συστηματικά η έλεγχη ε, της νομιμότητας στην δραστηριότητα των μελών. Ο κύριος Ιόγκο, πρόεδρε, δεν έχω για τη συγκεκριμένη υπόθεση του ελεγκτικού συνέδριου συγκεκριμένε Ευχαριστώ και ο Γενικός Γραμματεύς τώρα παρακαλώ για να απαντήσετε. Πρόεδρε, να ξεκινήσω από τα κοινωνικά δίκτυα. Στο Twitter έχουμε 17.500 ε, followers, 10.000 στο LinkedIn, στο YouTube 863 δεν έχω τα στοιχεία των προηγουμένων ετών αλλά θα τα αποστείλω στον κύριο Σαλαφράγκα και στην Επιτροπή. Στις προηγούμενες ερωτήσεις που υποβάλατε, στην 15, για τους υπαλλήλους ε, που ελάμβαναν αποζημιώσεις δεν είχαν λάβει κανένας τέτοιου είδους αποζημιώσεις. Είχαμε κάποιες περιπτώσεις συμμετοχής σε επιτροπές επιλογής ε, διαγωνισμών της ΕΠΣΟ και οι μόνες αποζημιώσεις που είχαν γίνει ήταν σχετικά με, τις, ε, με την ε, μεταφορά, με το ταξίδι και ενδεχομένως με κάποια διανυκτέρευση που χρειάστηκε να κάνουν. Για τα καθήκοντα που κεντρικοποιήσαμε στο Paymaster Office αυτό που κάναμε είναι ότι μεταφέραμε μια σειρά καθηκόντων την μισθοδοσία, τις αποστολές, δηλαδή καθήκοντα που δεν συνδέονται άμεσα με την ε, λειτουργία του οργάνου, γιατί είχαμε κεντρικοποιήσει κάποια, κάποιες υπηρεσίες ε, λογισμικού, και είναι το κεντρικό αυτό payment ε, office ε, που έχει αναλάβει αυτές τις κεντρικές λειτουργίες, το κάνουν και άλλα όργανα και λαμβάνει αμοιβή ανάλογα με τον αριθμό των φακέλων που λαμβάνει. Πριν από δύο χρόνια, για παράδειγμα, μεταφέραμε μία θέση και αυτό μας επέτρεψε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και να διατηρήσουμε τους, ε, το προσωπικό στους ελέγχους που βεβαίως είναι και το πιο σημαντικό πεδίο της ε, δραστηριότητά μας. Στην ερώτηση 37 το συνέδριο πρόσεξε ιδιαίτερα ε, την πιστοποίηση αυτή έμας που προϋποθέτει μια προπαρασκευή σημαντική προκειμένου να διατηρήσουμε τα πρότυπα και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Αν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία που χρειάζεστε, γιατί έχουμε μια λεπτομερέστατη έκθεση επί της πιστοποίησης μας, ε, που θα διαβάσουμε στην Επιτροπή, που δίνει λεπτομερείς πληροφορίες για όλους τους δείκτες και την αξιολόγηση. Αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μια νέα πρωτοβουλία για να μειώσουμε στο ελάχιστο ή, και να καταργήσουμε τελείως τη χρήση πλαστικών, λέει ο μιλητής. Νομίζω ότι και σε αυτό θα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα. Τώρα σε σχέση με, με τα έργα ασφάλεια, Secure Place Project, ήταν μία ενιαία και μοναδική δαπάνη σχετικά με την ε, ασφάλεια της περιμέτρου του συνεδρίου ώστε να υπάρχει μια περιοχή, ζώνη δηλαδή, πιστοποίηση και ελέγχου το οποίο έγινε μετά από έναν έλεγχο για την Ισπανική αστυνομία και με τη βοήθεια της αστυνομίας του Λουξεμβούργου και υποστήριξη από κάποιες μονάδες της Ιντερπολ, που είχαν διενεργήσει μελέτες και για άλλα έργα όπως και για το δικαστήριο εγκαταστήσαμε κάποιες κάμερες ασφαλείας και αυτό ήταν στην ουσία το σύστημα ασφάλειας στο οποίο προχωρήσαμε το έργο. Υπάρχει, υπάρχουν και κάποια πρόσθετα στοιχεία πρέπει ακόμα να ολοκληρωθούν όπως τα μεγάφωνα στο εσωτερικό των αιθουσών σχετικά με ειδοποίηση για έκτακτη ανάγκη, πυρκαγιέ κτλ. Αλλά και αυτά είναι στα πλαίσια μοναδικής και ενιαία δαπάνη. Για την συνεργασία με τους ομολόγους ε, του ελεκτικού συνεδρίου, αυτό ρυθμίζεται από τη συνθήκη, διενεργούμε τους ελέγχους μας ε, στην συντριπτική της πλειοψηφία στα κράτη-μέλη και γι' αυτό υπολογίζουμε και βασιζόμαστε στην πολύτιμη συνεργασία με τα συνέδρια των κρατών μελών. Υπάρχει μια, ένα συντονισμός αρκετά ρευστός, υπάρχει μια ετήσια συνάντηση συντονισμού μεταξύ των εκπροσώπων των ελεκτικών συνεδρίων και υπάρχουν και άλλες ε, επαφές και συναντήσεις ε, προκειμένου να υποστηρίξουν το δίκτυο αυτό για την ανταλλαγή πρακτικών, για τα προγράμματα κατάρτισης. Επίσης, έχουμε μια ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, ένα πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων με εθνικούς εμπειρογνώμονες ή με δικούς μας υπαλλήλους που συνεργάζονται με τις υπηρεσίες των κρατικών ελεκτικών συνεδριών, των κρατών μελών δηλαδή. Για την ερώτηση του κυρίου Γιάβορ για τον συστημικό ή όχι χαρακτήρα του ζητήματος, η έκθεση του Όλαφ δεν αναφέρεται σε κάποια συστημική ε, περίπτωση, αναφέρεται σε επιμέρους περίπτωση. Παρόλα αυτά, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Ελένε, διενεργείται ένας έλεγχος ε, σύγκρισης του, της λειτουργίας του παλαιού συστήματος και του υφισταμένου και νομίζω ότι θα μπορέσει εκείνος να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού όταν εμφανιστεί, όταν παρεστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ε, Γενική Γραμματέα για την ε, πληρότητα των απαντήσεών σας και την διασημότητα να απαντήσετε ερωτήσεις ε, πρόσθετες εφόσον υπάρξουν. Ας, ας προχωρήσουμε τώρα στα υπόλοιπα όργανα. Ίσως μπορούμε από κοινού αυτά να τα δούμε και ίσως ο κάθε Γενικός Γραμματέας ε, να έχει πέντε λεπτά στην ε, αρχική του τοποθέτηση. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ΕΟΚΕ. Ο κύριος Μπρουνέτη είναι ο Γενικός Γραμματέας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι το 2017 συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες μας με βάση και την νομοθετική μας εντολή. Η ΟΚΕΑ υιοθέτησε τις ε, εκθέσεις και συστάσεις της, ε, κάνει μεγαλύτερη προσπάθεια για την επικοινωνιακή της ε, πολιτική και την ανταπόκριση και σε τοπικό επίπεδο ενώσεις δηλαδή ε, εργοδοτών και ε, εργαζομένων και λοιπούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Μια σειρά από διαφορετικές δραστηριότητες που ονομάζονται going local αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα, συγκεκριμένε δράσεις δηλαδή, που αναπτύσσουν τα μέλη μας ε, στα κράτη-μέλη προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερη επικοινωνία και επαφή με τους διαφορούς παράγοντες και τα στοιχεία της κοινωνίας, συγκεκριμένα παραδείγματα για, παραδείγματα για τη συμβολή στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαβούλευση για τη Λευκή Βίβλο στο μέλλον, για το μέλλον της Ευρώπης με 27 διαφορετικές συζητήσεις που οργανώθηκαν στα κράτη-μέλη και συμμετοχή άνω των χιλίων συμμετεχόντων. Είχαμε επίσης συμμετοχή ενεργό στις δραστηριότητες τις σχετικές με το Ευρωπαϊκό ε, Εξάμεινο και τον Κοινωνικό Πυλώνα. Είχαμε επίσης σημαντικό στοιχείο την δημιουργία από εκείνο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Πλατφόρμας για την Κυκλική Οικονομία, ένα στοιχείο που ιδιαίτερα ενδιαφέρει την Επιτροπή μας, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται και στο επίκεντρο όλης νομοθετικής δουλειάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επικοινωνία επίσης έχουμε σημαντική αύξηση. Μέσω του Twitter 20% και του Facebook 24% της επικοινωνίας μας. Άρα Είμαστε κάπου στους 25.000 ε, με 30.000 χρήστες, για να απαντήσω στην ερώτηση του ερωτηματολογίου. 96,5% η απήχηση και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γιατί αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί και στην ε, αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία που ε, υιοθετούμε ιδιαίτερα αισθανόμαστε ικανοποιημένοι δε από το γεγονός ότι και το 2017 όπως και το παρελθόν δεν είχε ε, ειδικέ παρατηρήσεις στο ελεκτικό συνέδριο για, τις, ε, για την εκτέλεση του προπολογισμού μας. Προσωπικό 2017 προχωρήσαμε και ολοκληρώσαμε την κατά 1% ε, μείωση του προσωπικού όπως είχε αποφασιστεί από τη Διοργανική Συμφωνία του 2013 έτσι λοιπόν και με τις μεταφορές προσωπικού για το κέντρο έρευνας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μειώσαμε κατά 8,1% και 59 θέσεις στο προσωπικό μας. Επίσης, ιδιαίτερη η ικανοποίηση νομίζω ότι μπορούμε να εκφράσουμε και για τα συγκεκριμένα ε, νούμερα σε σχέση με την ισότητα των φύλων. 53% γυναίκες στο middle management, στη μέση διαχείριση 50% στην ανώτερη διαχείριση. Ε, συμφωνία του 2014 με το Ευρωπαϊκό 2013, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ε, συνεχίζεται και έχει να κάνει με την επαφή για διάφορα θέματα και σημεία επικοινωνίας ε, και πρωτοβουλίες ε, μεταξύ εισηγητών των, διαφορών, των δύο αυτών θεσμικών οργάνων αλλά, και με, οργάνων αλλά και με την Επιτροπή των Περιφερειών. 2017 μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση της Συμφωνίας Συνεργασίας μας δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα για κοινή χρήση των υπηρεσιών μετάφρασης της πληροφορικής των κτηρίων και της ασφάλειας ασφάλειας με σημαντικό και οικονομία κλίμακος. Για τον φορολογούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δύο στοιχεία που μας απασχολούν ακόμη και άλλο ένα τρίτο που θα εκθέσω προς το τέλος. Έχουμε η υποεπένδυση πάντα σημαντική ως προς την πληροφορική. 3% του προϋπολογισμού μας είναι οι σχετικές δαπάνες, ενώ τα μεγαλύτερα θεσμικά όργανα έχουν 7%. Ε, επενδύσεις και αυτό το καλύπτουμε με συστήματα ραμασάζ ε, στο τέλος του χρόνου. Επίσης, ε, ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί είναι τα κτίρια και οι αίθουσε συνεδριάσεων. Προσπαθούμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσουμε την χρήση του κτηρίου Βαρμέρλαντ που βρίσκεται σε μίσθωση αυτή τη στιγμή μαζί με την Επιτροπή των Περιφερειών όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λάβει τη σχετική απόφαση. Και επίσης, επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, να πω δύο λόγια για το πρόβλημα της παρενόχλησης. Ξέρω ότι κυκλοφορούν διάφοροι μύθοι και άρθρα. Θα ήθελα να πω πως ε, η ΟΚΕ με πολύ μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ε, παρενόχλησης και πρωτοβουλίες των μελών μας κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου και ενεργό συμμετοχή των Προέδρων των Ομάδων. Γίνεται μια μελέτη ένας δημόσιος διάλογος και αναλογισμός που θα πρέπει να ε, καταλήξει στην ενσωμάτωση ενός διοικητικού συστήματος εργαλείου ε, για την ε, αντιμετώπιση και πρόληψη της παρενόχλησης. απόφασίς έχουν ληφθεί χρόνια τώρα και έχουμε μία ε, θεσμική προσέγγιση με τον ε, ε, σύμβουλο από κρούο λοιπόν με τα ή οδήποτε υπενιγμό που θα οδηγούσε στο συμπέρασμα πως η διοίκηση δεν επιτρέπει στους υπαλλήλου να εκφράζονται ελεύθερα. Του αντίον οποιοδήποτε υποφέρει, έχει ζητήματα, δυσκολίες στον χώρο εργασίας του, καλείται να εκδηλώσει τις ε, σκέψεις του. Είχαμε ένα θέμα συγκεκριμένο και χωρίς να θέλω να δώσω λεπτομέρειες δεδομένου ότι πρόκειται για θέμα απορρίτου και πρέπει να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα του ε, ενδιαφερομένου, δεδομένου ότι έχουμε την υποχρέωση της ε, μέρημνας, δυνάμει και του σχετικού κανονισμού. Δεν αποκλείεται λοιπόν ε, καμία επιλογή ως προς την ε, μελέτη και εξέταση προβλημάτων που έχουν να κάνουν με την ψυχολογική, την ηθική, οποιαδήποτε άλλη μορφή παρενόχληση. Δεν έχουμε κανένα περιορισμό λοιπόν, γιατί έχουμε πάνω απ' όλα καθήκον να προστατεύουμε τους υπαλλήλους μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να πάμε τώρα στην Επιτροπή των Περιφερειών. Ο κύριος Μπούριεν, ο Γενικός Γραμματέας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θα είμαι πολύ σύντομος διότι είχαμε διατρέξει αρκετές ε, σημαντικές διοικητικές ε, λεπτομέρειες. Θα σας αναφέρω σχετικά με τρία ζητήματα. Το πρώτο είναι η προετοιμασία του έτους 2019 εκλογικός μιλώντας. Το δεύτερο είναι η συμφωνία συνεργασίας ε, με την ΕΟΚΕ, αλλά βεβαίως και με εσάς, τη συνεργασία δηλαδή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου φέτος μάλλον σε λίγο, το Φεβρουάριο του 19 θα έχουμε ολοκληρώσει μια πενταετία συνεργασίας και θα μου επιτρέψετε να σας ε, κάνω μια σύντομη ενημέρωση για την συνεργασία πέραν του παρόντος πλαισίου. Λοιπόν, τι κάναμε το 2017 για τις ευρωαϊκές εκλογές ε, του 19. Όπως ανέφερε πρόσφατα και ο πρόεδρος Ταγιάννη, το θέμα είναι ευρωπαϊκής και τοπικής δημοκρατία και με την ευκαιρία θα υπογράμμιζα τις διαθεσμικές συνέργειες που επιτύχαμε και σε πολιτικό και σε διοικητικό επίπεδο, δηλαδή των διευθύνσεων επικοινωνίας, στα πλαίσια των διαθεσμικών εκστρατιών, εμείς είμαστε πεπισμένος εταίρος της κοινή προσπάθειας που γίνεται και προάγουμε το θέμα μέσω των ε, εκδηλώσεων που διοργανώνουμε και μέσω των κοινωνικών δικτύων. Επίσης έχουμε συστηματικό διάλογο σε τοπικό επίπεδο με τις ε, πόλεις και τις περιφέρειες των μελών και με την υποστήριξη της ε, αρχής προϋπολογισμού διοργανώσαμε 180 διαβουλεύσεις πολιτών το 2017 επίσης αναπτύξαμε μια διαδικτυακή πύλη online που ήρθε σε επαφή με άνω των 40.000 πολιτών και ψηφοφόρων που τους υποστηρίζει στην άσκηση των δημοκρατικών τους καθηκόντων. Είχαμε και την Europe.com, την μεγαλύτερη εκδήλωση επικοινωνίας της Βρυξέλλες, προκειμένου να έχουμε μια πραγματικά πραγματική συμμαχία 1500 αποκεντρωμένων ε, υπευθύνων επικοινωνίας υποστηρίζοντας ε, το ευρωπαϊκό αυτό έργο και με διαγωνισμό που θα ακολουθήσει στους ερχόμενους μήνες. Θα ήθελα να αναφερθώ και στην ε, πολύ πετυχημένη συνεργασία στον τομέα της επικοινωνίας, στο ευρύτερο πλαίσιο της ε, συμφωνίας συνεργασίας μας, όπου, όπως είπα, το Φεβρουάριο θα ε, γιορτάσουμε τα πέντε χρόνια της. Για την πολιτική συνεργασία, οι εισηγητές, οι πολιτικές ομάδες και οι εξειδικεμένες επιτροπές αύξησαν την ποσότητα και την ποιότητα της δουλειάς τους, και συμφώνησαν σε έναν μακροπρόθεσμο ε, σχεδιασμό ώστε οι γνωμοδοτήσεις μας να είναι πιο επίκαιρες το οποίο ισχύει για το σύνολο του φάσματος ε, του πολιτικού και νομοθετικού και εν ώψη του ΠΔΠ με το αίτημα που υποστηρίζουμε για 1,3 και το οποίο έχει διαβιβαστεί και μέσω του Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών προς όλες τις περιφερειές για να έχουμε και μια ε, ισχυρή συμμαχία συνοχής που αυτή τη στιγμή έχει 8.000 υπογράφοντες εκλεγμένα μέλη επιτύχαμε να αναπτύξουμε μια στρατηγική αλληλεγγύης με τρεις κατηγορίες ε, περιφερειών που διατηρούνται. Τα περιφερειακά προγράμματα είναι θεμελιώδους σημασίας ε, όπως ε, γνωρίζετε και για τους ε, πολίτες διότι οι πολίτες διερωτώνται διαρκώς τι κάνει η Ευρώπη για αυτούς. Τα 24 μέλη του προσωπικού που ε, μεταφέρθηκαν στο EPRS είναι απόδειξη της λειτουργικής μας, επιχειρησιακής μας μάλλον δέσμευσης στο πρόγραμμα αυτό και πολύ σύντομα καθότι πλησιάζω προς το τέλος ε, της παρουσίασής μου. Θα θέλαμε από κοινού μαζί σας να αναλάβουμε μια νέα θέση στον διαθεσμικό διάλογο, στον ενισχυμένο τακτικό διάλογο με τους πολίτες ε, που θα είναι ωφέλιμος ε, και σε τοπικό επίπεδο και εν των εκλογών των ευρωπαϊκών Αυτό είναι το όραμά μας για το μέλλον, όπου προσβλέπουμε και τη συνέχιση της πολύτιμης συνεργασίας μας. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Um, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Διανιέλο, παρακαλώ, από τον διαμεσολαβητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μεγάλη τιμή που μπορώ να Απευθύνω το λόγο στην Επιτροπή σας εκ μέρους του Διαμεσολαβητή από τη στιγμή που, για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβα ως Γενική Γραμματέας, ε, δίπλα μου ο κύριος για τα θέματα του προσωπικού και τα οικονομικά. Θα ήθελα να σας ενημερώσω καταρχάς για τις εξελίξεις που αφορούν τις κύριες δραστηριότητές μας, οι οποίες διαρκώς επεκτείνονται και στη συνέχεια να περάσω σε εσωτερικά ζητήματα, εκεί όπου προσπαθούμε δηλαδή να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και την ε, αποδοτικότητα των υπηρεσιών μας. Οι κύριες δραστηριότητες μας το 2017 συνεχίζονται με την εφαρμογή της στρατηγικής ε, του Ombudsman της Δημοσιογραφήτριας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας αλλά και της ορατότητας των εργασιών της υπηρεσίας μας για τον Ευρωπαίο πολίτη και ιδιαίτερα το δικαίωμα της αποκατάστασης ζημίας σε περίπτωση ε, διαχείριση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση Ως προς, την ορατότητα το 2017 σημειώνουμε συνεχή ε, και σταθερή ανάπτυξη, αύξηση του αριθμού των μελών, κυρίως στο Twitter και στο Instagram ε, των λογαριασμών μας. Γνωρίζουμε βεβαίως ποια είναι τα όρια των δυνατοτήτων μας και γι' αυτό κάνουμε ιδιαίτερη ε, προσπάθεια για να στοχεύσουμε τους πολυπλασιαστές, αυτούς που θα μας βοηθήσουν δηλαδή να πλησιάσουμε ευρύτερο κοινό, ευρύτερα κοινά. Επίσης, για την ενίσχυση της ορατότητας ε, και σημειώνω ότι έχουμε λάβει ακόμη περισσότερες ε, διαμαρτυρίες από πολίτες στο ίδιο διάστημα του 2017 και άρα έχουν ανοίξει περισσότερες έρευνες. Ε, με όλο και μεγαλύτερο φάσμα. Τρία παραδείγματα θα σας δώσω, τα θεωρώ δηλαδή ε, αντιπροσωπευτικά του αντικτύπου, που επιδιώκουμε άλλωστε να εξασφαλίσουμε για τις δραστηριότητε του Ombudsman. Ε, το πρόβλημα των μη αμοιβόμενων ασκήσεων, πρακτικών ασκήσεων που αναφέρθηκε και νωρίτερα ήταν ένα θέμα που άνοιξε από νεαρό ή νεαρή Αυστριακή Επίσης, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τις γλώσσες ε, στις δημόσιες διαβουλεύσεις. Παράπονο που διατύπωσε ε, Ισπανός πολίτης η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων και ο ρόλος της ως προς την χορήγηση αδειών ε, εμπορευματοποίησης για διάφορες ποικιλίε καλαμποκιού αραβοσίτου κατόπιν παραπονού Γάλλου Όλα αυτά λοιπόν που είναι πολύ σημαντικά ζητήματα και θα ήθελα εδώ να αναφέρω πάλι στρατηγικές έρευνες που κάνουμε, που επίσης είναι πολύ σημαντικές. Ε, νομοθετικό έργο, πρόσβαση νομοθετικού έργου του Συμβουλίου, πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε ε, ιστοσελίδα και εργαλεία διαγραμμικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπηρεσία φαρμάκων και ο τρόπος με τον οποίο ασχολείται ή αντιμετωπίζει τους διαφορούς ε, τις διάφορες εταιρείε που αναπτύσσουν νέα φάρμακα πριν από την κίνηση της διαδικασίας, δηλαδή το pre-submission activity όπως ονομάζεται, η συνολική συμμόρφωση ε, στις συστάσεις του, της Ombudsman ή στις προτινόμενες λύσεις ήταν σε επίπεδο ευρωπαϊκών οργανών 85%. Στα δε εσωτερικά ζητήματα και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας μας, γιατί θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο αυτό προκειμένου να, ενισχυθεί η δυνατότητα επέκτασης των κύριων ε, δραστηριοτήτων μας. Θα ήθελα καταρχάς να σημειώσω με ικανοποίηση πως το 2017 μπορέσαμε να τηρήσουμε το ποσοστό της στήριξης του προπολογισμού μας στο 95%. Δεύτερον, η ε, διαμεσολαβήτρια υιοθέτησε μια συνολική πολιτική, ένα πλαίσιο πολιτικής ε, για το 2017 γενικά για το προσωπικό και αρχίσει να αναπτύσσει μια σειρά από συναφείς πολιτικές. Επιτρέψτε μου λοιπόν ιδιαίτερος να τονίσω την πολιτική για την πρόληψη και προστασία κατά της παρενόχλησης όπου σαφώς αναφέρεται μηδενική ανοχή, προσέγγιση μηδενικής ανοχής από την Ομπουτσμαν για κάθε μορφή παρενόχληση. Το 2018 αυτό οδήγησε στη θέσπιση του ε, ε, Συμβούλου του θεσμού του Συμβούλου Δεοντολογίας αλλά και μια σειρά από προτάσεις για την πρόληψη και προστασία από την παρενόχληση ιδιαίτερα με την υποχρεωτική κατάρτιση όλων των στελεχών στην οποία αναποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία. Ε, επίσης, η Διαμεσολαβούτρια ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στην ισότιμη αντιμετώπιση των φύλων, ε, πράγμα το οποίο θεωρεί πως έχει επιτευχθεί επιτυχώς και στις θέσεις ε, διαχείρισης και στο γενικό διοικητικό προσωπικό. Επίσης και πολύ σημαντικό, θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω την βελτιωμένη αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των ε, διαμαρτυριών και προσφυγών των πολιτών, που είναι κύρια, των κύριων καθήκων μας, με σημαντική βελτίωση από το 2016. Έχουμε μπορέσει να δίνουμε απαντήσεις ε, πιο έγκαιρες ε, στους πολίτες πράγμα το οποίο ήταν σοβαρό στόχος ε, της ε, υπηρεσίας μας. Έχει μειωθεί από τις 340 ημέρες το 2016 στις 266 ημέρες ως χρόνος ανταπόκρισης το 2017. Το 2017 μπορέσαμε να κλείσουμε 57% του συνόλου των ερευνών μας μέσα σε ένα εξάμεινο. 87% μέσα σε 18 μήνες, κάτι το οποίο ξεπέρνασε τον, τους κύριους δείκτες και στόχους που είχαμε για τις δύο αυτές κατηγορίες ε, αντίστοιχα κλεισίματος ερευνών και η θετική τάση συνεχίζεται ε, και το 2018. Εν τέλει το Φεβρουάριο του 2018 και ύστερα από μια δοκιμαστική περίοδο που ξεκίνησε προς τα τέλη του 2017 ε, κινήσαμε Επίσημώ στην ε, διαδικασία ταχεία πρόσβαση, ταχεία ολοκλήρωσης ως προ την πρόσβαση σε ε, έγγραφα θεσμικών οργάνων ε, προκειμένου να διευκολυνθεί αυτό. Είναι μια δοκιμαστική φάση που ύστερα από ένα χρόνο εκτέλεσης θα αξιολογηθεί και κλείνοντα θα ήθελα δρατώμενη τη ευκαιρία που μου δίνετε να ενημερώσω την Επιτροπή σα για τη θετική εμπειρία που είχαμε και από την απονομή του βραβείου για την βέλτιστη ε, διοικητική πρακτική και έτσι επαναλήφθη και για φέτος αυτή η διαδικασία. Έχει ανοίξει τώρα, εδώ και ένα μήνα. Είναι ανοιχτές οι υποψηφιότητες ακόμη. Ελπίζουμε να λάβουμε πολλές υποψηφιότητες από όλα τα θεσμικά όργανα και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νάβας ε, τελευταίος, αλλά εξίσου μηχανή, ε, σημαντικός από τον επόπτη προστασίας δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω εκ μέρους του υπόπτη δεδομένων. Μαρίνα Σάντσεθ Λόπες ε, είναι η αντίστοιχη τμήματάρση που είναι δίπλα μου και θα ήθελα να πω ότι χάρη στη δική της ομάδα είναι τα του οίκου μας εντάξει. Είμαστε το πιο μικρό θεσμικό όργανο. Θα προσπαθήσω να είμαι και πιο σύντομος λοιπόν από τους προηγούμενους εγώ σήμερα στην παρέμβασή μου, διότι είναι μια μικρή υπηρεσία μεν, όχι όμως ότι και δεν παίρνουμε σοβαρά υπόψη τις οικονομικές μας υποχρεώσεις. Προσπαθούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του οργανισμού μας. Τρία πράγματα κάνουμε. Υποπτεύουμε τη διαδικασία προσωπικών δεδομένων από τις ε, ευρωπαϊκά όργανα για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει μια καλή κουλτούρα προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Και εμείς πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα Χρησιμοποιούμε λοιπόν και τα μέσα που μας προσφέρει ο νέος κανονισμός ε, και συγκεκριμένα 11 Δεκεμβρίου ε, θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις δυνατότητες αυτού του νέου κανονισμού για να δώσουμε όθηση στην προστασία των δεδομένων. Επίσης παρέχουμε συμβουλές στον αρμόδιο. Οι 28 διαβουλεύσεις λάβαμε το 18 και για το 19 έχουμε ήδη λάβει 61 Τέλος, από το Μάιο του 2018 παρέχουμε και γραμματική υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων που δημιουργήθηκε μετά από την θέση ισχύ του Γενικού Κανόνισμου Δεδομένων. Το 2017 ήταν μια μεταβατική χρονιά σκληρή δουλειά κάναμε. Ξεκινήσαμε με την εποπτεία της Europol, του Ευρωπαϊκού FBI δηλαδή, Προετοιμαστήκαμε για την δημιουργία του νέου νομικού πλαισίου και επίσης έχουμε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πλέον ε, θεσπίσει, που είναι ένα μεγάλο βρήμα για το μικρό μας οργανισμό. Από τις πληροφορίες που σας στείλαμε θα δείτε ότι όλες τις στάσεις του 16 της απαλλαγές έχουμε εφαρμόσει και κλείσαμε ή θα κλείσουμε, τόσο πάντων μέχρι τα τέλη του έτους, ε, όλες τις συστάσεις ε, των εσωτερικών ελεγκτών. Άρα Συμπεραίνω λέγοντας αυτό που είπα ουσιαστικά και στην αρχή. Ότι παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη ευθύνε μας και είμαστε υπερήφανοι ότι για 7η συναπτή χρονιά η διασφάλιση, η δήλωση διασφάλιση 17 του Ελεκτικού Συνδέρου δεν περιέχει καμία παρατήρηση σε ό,τι αφορά του ετήσιου μα λογαριασμού και την ετήσια έκθεση πεπραγμένου. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και παραμένω στην διάθεση σα για ερωτήσει. Ευχαριστούμε. Να πάμε τώρα στην ε, εισηγήτρια, την κυρία Γιαλασέντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις. Στην περίπτωση της ΕΟΚΕ, να συγχαρώ τον κύριο Μπρουνέτη γιατί μόλις ορίστηκε 14 Νοεμβρίου νέος Γενικός Γραμματέας ήθελα να ρωτήσω, να τον ρωτήσω, καθότι ήταν ε, προηγουμένως ε, προϊστάμενος ανθρωπίνων πόρων και προϋπολογισμού, πότε έχει σκεφτεί να ορίσει το νέο Γενικό Διευθυντή ακριβώς ανθρωπίνων πόρων και προϋπολογισμού στη θέση του. Δεύτερον, να τον ευχαριστήσω για τον καλό συντονισμό που διατηρήθηκε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου είχαμε και κάποιους ε, συγκεκριμένους φακέλους πολύ ενδιαφέροντες ε, κοινωνικά, με σημαντικό δηλαδή αντίκτυπο, όπως και με την Επιτροπή των Περιφερειών, κατόπιν συστάσεως βεβαίως αυτού του Κοινοβουλίου. Τώρα εγώ εδρώ εξ ονόματος του κυρίου Κον ε, και από τον οποίο προέρχεται η ερώτηση σχετικά με τις δαπάνες για το σύστημα του λογισμικού που του φαίνεται κάπως ε, χαμηλό το επίπεδο αυτό. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια αλλαγή ή κάτι που, ε, στο οποίο θα μπορούσαμε εμείς να βοηθήσουμε επ' αυτού. γιατί το να ε, περιορίζουμε, να στραγγαλίζουμε δηλαδή ε, τις δαπάνες ε, καμιά φορά αυτή η υποχρεωτική πίεση προς τα κάτω οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερα τελικά έξοδα. Τώρα, είχαν βελτιωθεί πάρα πολύ τα θέματα της συνεργασίας με όλη τη συμφωνία για το κόστος των αποστολών, τα βιογραφικά. Ε, σας συγχαίρω για όλα αυτά και σας ευχαριστώ. Βλέπουμε ότι το κόστος των αποστολών μειώθηκε κατά 19 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο μας φαίνεται εντυπωσιακό. Και αν θέλει ο κύριος Μπρουνέτη να σχολιάσει κάτι περαιτέρω επ' αυτού, ας το κάνει. Τώρα, ο εσωτερικός κανονισμός και ο κώδικας διοντολογίας δεν τα μέλη, στην απάντηση δηλαδή 51, μας οδηγεί σε μια παρατήρηση. Καθότι έχετε αρχίσει να διανέμετε κάποια στοιχεία περιπτώσεων κρουσμάτων παρενόχλησης θα ήθελα να μας εξηγήσετε με σαφήνεια με ποιο τρόπο σκοπεύετε να ενημερώσετε ή να ευαισθητοποιήσετε τα μέλη της Επιτροπής σας που προέρχονται από τελείως διαφορετικά περιβάλλοντα σχετικά με την περιοδική εμφάνιση, τέλος πάντων την παροδική εμφάνιση τέτοιων κρουσμάτων προκειμένου να αναπτυχθεί μία εν πάση περιπτώσει προσέγγιση διοικητική ως προς το θέμα αυτό. Για την ε, ερώτηση 47 μας λέτε από ό,τι φαίνεται ότι καμία περίπτωση δεν οδηγήθηκε στον Όλαφ αλλά εμείς είχαμε μια επιστολή λάβει από, τις, από τα συνδικάτα που φαίνεται ότι από ό,τι φαίνεται υπάρχουν τέσσερις περιπτώσεις υπό εξέταση αυτή τη στιγμή στον Όλαφο, οπότε θα ήθελα να μας το εξηγήσετε αυτό. Ε, ως προς την ε, προσφορά και την χρήση των ε, ευέλικτων μέσων εργασίας, φαίνεται ότι είναι οι γυναίκες που το ζητούν αυτό και ε, ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον τους πατέρες που, είναι και, που συνεργάζονται, που είναι μέλη του προσωπικού σας, εάν τους ε, προσφέρετε κάποιες ε, δυνατότητες στο πλαίσιο αυτό. Τώρα, είχαμε πολύ σε διμερείς επαφές ε, με την Επιτροπή και ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη συνεργασία. Να ρωτήσω εάν εξακολουθείτε να έχετε μία Ε, συνεχιζόμενη ανταλλαγή με το EPRS ε, σχετικά με το προσωπικό, αν αυτό δηλαδή συνεχίζεται ή αν έχετε καταλήξει σε μια τελική συμφωνία. Από την άλλη, στα θέματα ε, φίλων τα πράγματα επιδεινώνονται. δεν βλέπουμε περισσότερες, αλλά λιγότερες θέσεις σε ανώτερες διοικητικές, γυναίκες με συγχωρείτε σε ανώτερες διοικητικές θέσεις. Ήθελα να ρωτήσω αν αυτό οφείλεται στην συνολική μείωση των υπαλλήλων ή τι άλλο, με τι άλλο σχετίζεται και τέλος θα θέλαμε να καταλάβουμε πώς θα εφαρμοστεί η απόφαση του δικαστηρίου του Οκτωβρίου 18 για τον ε, προηγούμενο ελεγκτή. Πώς σκοπεύει να υλοποιήσει το σχετικό, την απόφαση αυτή ο κύριος Μπρουνέτη. Για τον διαμεσολαβητή να ευχαριστήσω. Έχουμε εδώ μια ε, γενική γραμματέα την οποία καλωσορίζουμε. Βλέπουμε ότι η επιφάνεια των δηλώσεων και των παρεμβάσεων του διαμεσολαβητή είναι όλο και πιο σημαντική. Επίσης ε, είχαμε μια σημαντική αύξηση του flexi-time και της τηλεεργασίας στην υπηρεσία και θέλαμε να ρωτήσουμε κατά πόσο αν έχετε προχωρήσει μια αξιολόγηση αυτών των διευθετήσεων και τι θα είχατε να συστήσετε από αυτού σε άλλα θεσμικά όργανα. Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον της, ε, την έρευνα για την προσβασιμότητα στους χώρους της Επιτροπής και την διαφάνεια των ε, διαπραγματεύσεων για τον Brexit. Έχουμε επίσης σημαντική αύξηση ε, συμβασιούχων και προσωρινών, το οποίο σημαίνει ε, ιδιαίτερα στην περίπτωση των σταζιέρ, σας ρωτώ αν αυτό απορρέει από τη μείωση του προσωπικού, γιατί δεν μας φαίνεται ότι προχωρούμε εδώ προς την σωστή κατεύθυνση. Για τον επόπτη, ε, προστασίας δομένων, βλέπουμε, και το θεωρώ αυτό θετικό στοιχείο, μια αύξηση 21% του προϋπολογισμού ακριβώς λόγω της νέας εντολής ε, για τη νέα νομοθεσία, δηλαδή προστασίας δεδομένων όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται και είναι σημαντικό αυτό, έχει παγκόσμιο αντίκτυπο αλλά θέλαμε να κατανοήσουμε ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουν αυξηθεί στα πλαίσια αυτής της νέας εντολής. Ο επόπτης υποστήριξε και την ε, δημιουργία της ε- Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προστασίας των Δεδομένων και θέλαμε να καταλάβουμε ποια θα είναι τα καθήκοντά της, οι αρμοδιότητες της, σε σχέση με τον επόπτη και επίσης να αναφερθώ στον κατάλογο για τη διαφάνεια των αποστολών, των διαγωνισμών. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank move. Ευχαριστώ να περάσουμε στους και όλες τις και λοιπούς συναδέλφους που ενδεχομένω θέλουν ε, το λόγο. Πρώτα απ' όλα για δύο λεπτά καιρός, αλλά Αλαφράγκα τα καλύψτε όλους, έτσι ναι. Ε, πράγματι, σε ό,τι αφορά την ΕΟΚΕ και την Επιτροπή των Περιφερειών, είχαμε πολλές εκθέσεις και συναντήσεις, ενισχύθηκε η συνεργασία ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα όμως να κάνω κάποιες ερωτήσεις για να διευκρινιστούν ορισμένα πράγματα. Σε ό,τι αφορά τη χρήση του προπολογισμού στην ΕΟΚΕ βλέπουμε μείωση από το 97,2 το 2016 το 96,1 για το 17. Εξήγηση υπάρχει. Απάντηση στην ερώτηση 10 για τον αντίκτυπο που μπορούσε να έχει το Brexit. Δεν μας δίνεται νούμερα και είναι αόριστη απάντηση. Νομίζω θα ήταν σχετικά εύκολο να μας δώσετε κάποια νούμερα για το κόστος των ε, ταξιδίων, τα οδηπορικά των βετανών μελών. Για το 23, σε ό,τι αφορά τις παθήσεις burnout, δεν απαντάτε παρκώς. Υψηλά επίπεδα στρες, οι άδειε λόγω του στρες, φαντάζομαι ότι έχουν κάποιο πιστοτικό ιατρικό. Και σε ό,τι αφορά την ενεργική απόδοση και το κόστος μίσθωσης για τις δύο συμβουλευτικέ επιτροπές. Δίνετε τα στοιχεία από κοινού και όχι χωριστά. Δεν ξέρω, σε ενεργειακή απόδοση εντάξει, αλλά για το ενίκιο νομίζω ότι μπορούμε να τα πούμε διαφορετικά. Να δώσετε ξεχωριστά τα στοιχεία για τη διαμεσολαβήτρια, 29, για το εντελεργασία. Υπάρχει διάκριση που θα μπορούσε να γίνει των δεδομένων μεταξύ ανδρών και γυναικών μα δίνετε εναρμονισμένη απάντηση. Θα ήθελα κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία και σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασία Δεδομένων, μα λέτε ότι δεν έχετε τεχνικά μέσα για να αναφέρετε τις ασθένειες. Δεν υπάρχουν στατιστικά. Στην 20 ερώτηση λέτε ότι γίνεται αυτό με το χέρι και προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο σύστημα της Κομισιόν. Τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε για να έχετε πρόσβαση στο σύστημα της Κομισιόν Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριος Κλίντ είναι ο επόμενος. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την ΕΟΚΕ. Ε, είχα μια ερώτηση που την έβαλε ο συνάδελφος Χαβιέρα, άρα να μην επαναλάβω. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή των Περιφερειών, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις ε, της αποχώρησης ε, της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας δίνεται ένα νούμερο για το 2019 γύρω στα 300 τόσα χιλιάδες και γύρω στα 500 τόσα για το 2019. Πώς ε, φτάνετε σε αυτά τα νούμερα. Επίσης, ε, τι γίνεται με τις εργασιακές ε, συνθήκες στις, στην Επιτροπή των Περιφερειών. Υπάρχει μια αρνητική εκτίμηση σχετικά. Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις και υπάρχει η περίπτωση Ρόμπερτ Μακόη που ήταν συνεργάτης ε, της Επιτροπής έχει φύγει εδώ και χρόνια κατόπιν πιέσεων και υπήρξαν διάφορες καταγγελίες ε, και πρόσφατα φέτος ο Μακόη πήγε, τρεις, ε, πήγε στο δικαστήριο και κέρδισε για τρίτη φορά. Παρόλα αυτά δεν είναι διατεθειμένη η Επιτροπή των Περιφερειών να, να δεχθεί ε, την ετοιμιγορία του δικαστηρίου και να ζητήσει συγγνώμη από τον ε, υπάλληλο αυτό. Θα με ενδιέφερε η τελευταία ε, τη λέει της ε, Επιτροπής των Περιφέρειων σε ό,τι αφορά το διαμεσολαβητή γίνεται για κάποια ταξίδια πόσο συχνά γίνονται τέτοια ταξίδια διερευνητικά και αν έχετε κάποια στοιχεία να μας δώσετε. Επίσης ότι αφορά ε, το ποσό των 60.000 που ανέφερε επόπτης για εξοπλισμό. Τι ε, εξοπλισμός είναι αυτός και πώς κατανέμεται. Ευχαριστώ. Επόμενος ο κ. Ντεγιόγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ένα διαδικαστικό. Θα ήθελα να παρακαλέσω η γραμματεία να γράψει ε, και να σημειώσει ότι θα ήθελα να συζητήσουμε τα περί απαλλαγής ε, στις εδρές των συντονιστών. Δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε ερωτήσεις και να πούμε σε βάθος και αυτό δεν είναι σωστό. Εγώ θα περιοριστώ στις δύο συμβουλευτικές επιτροπές, Επιτροπή Περιφερειών και ΕΟΚΕ για δύο πτυχές, από τη μία η διαφάνεια ορατότητα και από την άλλη η αποτελεσματικότητα. Σε ό,τι αφορά την ορατότητα, την προβολή, ε, πολύ καλή διάθεση και ενέργεια βλέπω να είστε πιο ορατοί. Όμως έχω κάποιες ερωτήσεις. Ίσως γραπτός, θα ήθελα να μου δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για τις τοπικές δραστηριότητες της ΕΟΚΕ και τι κάνει και η ΕΟΚΕ αλλά και η Επιτροπή των Περιφερειών για να προσφέρει κάποια πράγματα στους επισκέπτες που έρχονται εδώ στις Βρυξέλλες. Το Κοινοβούλιο ε, είναι ένας τουριστικός ε, προορισμός όλο και περισσότερο. Έχουμε το παρλαμεντάριο και άλλα ε, πράγματα που ενδιαφέρονται για τους. Τι κάνετε εσείς, οι δύο συμβουλευτικές επιτροπές, για να γίνετε και αυτό για να γίνετε και εσείς ελκυστικές εδώ στις Βρυξέλλες και να σας επισκέπτονται τουρίστες. Επιτροπή των 180 ε, διάλογοι σε πάνω από 110 περιφέρειες. Ταυμαστικό. Πολύ ωραία και πολύ καλά. Αλλά ποιος τα οργάνωσε, η Κομισιόν. Ποια ήταν προσθεμένη αξία από την Επιτροπή των Περιφερειών και αν όχι να μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες, αυτές που είχαμε λάβει γραπτός. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα, βλέπουμε η ΕΟΚΕ από τη μία έχει δείκτες, ε, βασικούς δείκτες ε, απόδοσης. Αυτό δεν το βλέπουμε στην Επιτροπή των Περιφερειών. Λέει ότι έχουμε διοικητικές δραστηριότητες και δεν μπορούμε να έχουμε δείκτες επιδόσεων. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά και συγκεκριμένα θέλω να πείτε ποιοι είναι αυτοί οι νέοι δείκτες που προβάλλει η ΕΟΚΕ. Okay. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Πρωτού ξαναδώσω το λόγο στους γενικούς γραμματείς. Μία πρόσθετη ερώτηση από μένα, μάλλον προς την Επιτροπή των Περιφερειών και την ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, σχετικά με το θέμα που οι συνάδελφοι έθεσαν αρκετές φορές, που είναι το Brexit. Θέμα το οποίο βεβαίως τον τελευταίο καιρό και τις τελευταίες μέρες σκεφτόμαστε πολύ Ποιε είναι οι σκέψει σα για τι μελλοντικέ σχέσει με το Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει ιδιαίτερα σε επίπεδο τοπικών αρχών, αποκεντρωμένων δηλαδή αρχών και κοινωνία των πολιτών. Έχετε ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση διατήρηση σχέσεων. Ε, επανέρχομαι τώρα στου Γενικού Γραμματεί για απαντήσεις. Παρακαλώ, η ΕΟΚΕ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να δώσω απάντηση στις ερωτήσεις, αν τυχόν. Μου ξεφύγει κάτι, σας το συγγνώμη τον προτέρων και Ευχαριστώ πολύ την κυρία για τα Σέντερ για τα ευγενικά της λόγια. Ένα σχόλιο που ακούστηκε σε σχέση με το μείωση των θαπανών ε, ταξιδιών και διαμονής των ε, μελών μας. Την απάντηση την έχουμε δώσει εάν κάνουμε την προσθήκη των εξόδων ε, κινήσεως και διαμονής των μετών μας, μείωση υπάρχει στο σύνολο, αλλά δεν είναι τεράστια. Επίσης, το ζήτημα της, ε, των υπεροεπενδύσεων στα θέματα της πληροφορικής, πώς μπορούμε να καλύψουμε το κενό. Μας έχει απασχολήσει και μας αυτό. Έχουμε κάνει σχετικές προτάσεις για το 2017 στα μέλη, αλλά ε, δεν έγιναν δεκτές. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να λάβουμε την άδεια της χρήσης ε, μόνο του προϋπολογισμού μας που δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί προς το τέλος του έτους για να βελτιώσουμε αυτή, αυτό το ποσοστό επενδύσεων στην πληροφορική. Για την ε, παρενόχληση και την πρόληψη, καλύτερα μια θετική εκστρατεία καταπολέμησης αυτής όπως είπα, είναι σε εξέλιξη σε επίπεδο κανονιστικό, διοικητικό ε, η εξετάση του θέματος. Ταυτόχρονα όμως ε, εξετάζουμε και την δυνατότητα ανάπτυξης μιας εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που έχει να κάνει με ε, μια καλύτερη αντίληψη της πολυπολιτισμικής, ε, του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος εργασίας για όλους μας. Αυτό απευθύνεται και στα μέλη και θα έχουμε οπωσδήποτε πολύ καλύτερη ανάπτυξη του προγράμματος του 2020 με την ανέωση των μελών. Όλαφ. Στην απαλλαγή ε, αναφέρεται ρητά ο όρος παρενόχληση στην απαλλαγή του 2017. Για το 2018 σας το είπα ήδη, δεν έχουμε κάποια καταγγελία παρενόχλησης. Αλλά βεβαίως παρακολουθούμε ενεργά και είμαστε στη θέση ή ουδήποτε εξωτερικού οργανισμού θελήσει να έρθει και να ελέγξει τη λειτουργία του, ε, της ε, ΕΟΚΕ. Επίσης, το ποσοστό συμμετοχής μας ρωτάτε, πώς μπορεί να ενισχυθεί το ποσοστό συμμετοχής των αρένων εργαζομένων ως προς μια πιο ευέλικτη μορφή εργασίας. Εάν ε, ωστόσο είναι λίγοι άντρες που εκμεταλλεύονται το σύστημα αυτό των ευέλικτων μορφών εργασίας, ε, πρέπει να πω ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι έχουμε πολλές γυναίκες στο προσωπικό μας. Δύο τρίτα είναι οι γυναίκες και άρα και εξηγείται, έτσι εξηγείται και η διαφορά. Η συγκέντρωση. Ε, καθηκόντων ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Διοικητικά είναι κάπως δύσκολο, αλλά θα γίνει. Κύριε Σαλαφράγκα. Ο κύριος Αλαφράνκα έθεσε το ερώτημα του χαμηλού ποσοστού εκτέλεσης. Κάποιες δραστηριότητες ε, ακυρώθηκαν πέρσι και έτσι εξηγείται σε ένα βαθμό αυτό το χαμηλό ποσοστό. Θεωρούμε όμως ότι δεν έχουμε πολύ, κακά, πολύ κακές επιδόσεις στην εκτέλεση. Το παρακολουθούμε όμως ότι βεβαίως θέλουμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με τα ποσά που μας διαθέτει η αρμόδια για τον προπολογισμό αρχή. Brexit. Οι πληροφορίες δεν είχαν περιληφθεί στο ερωτηματολόγιο. Να σας ενημερώσω για τα εξή. Θεωρούμε και άλλωστε ζητήσαμε και από την ε, αρμόδια για τον προπολογισμό αρχή να λάβει υπόψη αυτή την ε, πρόταση, ότι θα έχουμε 320 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα, γιατί πρώτον θα έχουμε 24, λιγότερους, 24 ε, λιγότερα μέλη, τους Βρετανούς δηλαδή πρώτο, δεύτερο, τρίτο εξάμεινο του 2019 και άρα το κόστος, οι δαπάνες συμμετοχής στις Ολομέλειες και στις, ε, στα θα μειωθούν. Επίσης, η αποζημίωση για τη χρήση της πληροφορικής που προβλέπετε για τα μέλη μας. Επίσης, ε, διαγράφεται για τα εν λόγω μέλη και τα τρία εξάμηνα του 19. Ε, η εξάντληση, burnout των εργαζομένων μας απασχολεί πολύ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει και σαν σύλληψη να αντιμετωπίσουμε και αυτό αφορά όχι μόνο εμάς αλλά και τις ιατρικές Μα υπηρεσίε, γιατί δεν αναγνωρίζεται σε ένα ιατρικό πιστοποιητικό η έννοια του burnout. Κάνουμε όμω μεγάλη προσπάθεια, φέρνουμε και εμπειρογνώμονες ε, για να μιλήσουν και με το προσωπικό που κινδυνεύει περισσότερο για να τους βοηθήσει ε, να διαγνώσουν τον κίνδυνο και ψυχοκοινωνικά βέβαια ε, και ξεκινούμε μια νέα μελέτη για να έχουμε δεδομένα πιο συγκεκριμένα για το θέμα αυτό που έχει τόσο μεγάλη σημασία. Ο κύριος De Jong ρωτάει για το οι δραστηριότητες going local. Θα σας προτείνω ε, να σας αποστείλουμε, να επιτρέψετε να σας αποστείλουμε γραπτές ε, απαντήσεις κύριε De Jong. Νομίζω ότι έτσι και χρόνια θα κερδίσουμε και πιο ικανοποιητικές ήταν οι απαντήσεις μας. Ε, ορατότητα, Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν εκδηλώσεις όπως η Μέρα της Ευρώπης ή άλλες, και νομίζω ότι εκπροσωπώ εδώ και την Επιτροπή των Περιφερειών, οι επιτροπές, οι δύο συμβουλευτικές επιτροπές, είναι μέσα στη διαδρομή. Από την πλατεία Λουξεμβούργου μέχρι το, η πλατεία Σούμαν έχουμε μια διαδρομή και εκεί βρισκόμαστε εμείς. Έχουμε κέντρο υποδοχής επισκεφτών στην Οδό Βελμπελιάρ με 8.000 κάθε χρόνο επισκέπτες. επομένω, νομίζω ότι έχουμε καλές επιδόσεις. Και επίση, κύριε Πρόεδρε, εσείς ρωτήσατε για το θέμα των σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, εάν μετά τι 29 Μαρτίου του 2019 και πάψει το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι μπορεί να συμβεί. Ε, μας έχει απασχολήσει λοιπόν το θέμα αυτό και σε όρους πολιτικούς. Έχω μια ομάδα εργασίας η οποία ασχολείται περισσότερο και με τις διοικητικές προστροπτυχές αλλά και με το μέλλον του φορέα μας και πιστεύω, χωρίς να θέλω βεβαίω να προδικάσω τι είδου αποφάσει θα ληφθούν σε πολιτικό επίπεδο, ότι σαφή είναι η βούληση για ανάπτυξη εγκαθίδρυση ενός πολύ στενού διαλόγου με τις αντίστοιχες αρχές του Ρωμένου Βασιλείου. Okay, um, I've got one item after this, where ε, έχουμε άλλο ένα σημείο και πρέπει να επιταχύνουμε. Ε, θα ζητούσα από τους υπόλοιπους ε, πέντε λεπτά, παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για την κυρία Γιάλα Σέντερ. Έχουμε σταματήσει με τις προσλήψεις έχουμε 24 υπαλλήλου σε ισοδυναμία με το EPRS. Επίσης, σχετικά με τους αναπληρωτές γενικούς διευθυντές και προϊσταμένους ε, τμήματων, ε, έχουμε προχωρήσει σε διάφορα πράγματα ενημέρωσης αλλά παρακολουθούμε τους μέσους όρους των υπολείπων θεσμικών οργάνων εκεί που υπολοιπόμαστε είναι στις ανώτατες ε, θέσεις λόγω του μεγέθους μας αλλά για το functional management είμαστε πάνω του 50% επομένως είναι αρκετά θετικό μέγεθος. επίσης λόγω οργανωτικών αλλαγών και κάποιων ε, ε, συμβάσεων ασφαλείας ε, προσφέραμε πιο μακροπρόθεσμες συμβάσεις σε κάποιο προσωπικό προσωρινής δηλαδή απασχόλησης. Τώρα, να πω ότι όπως και στην περίπτωση προηγουμένων αποφάσεων θα εφαρμόσουμε απολύτως τις αποφάσεις του δικαστηρίου και μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι έχουμε σαφέστατη πρόθεση να ε, κλείσουμε την συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία αναφερθήκατε και ε, προσυμμόρφωση ε, με τον κανονισμό του προσωπικού. Έχοντας εξετάσει προσεκτικά την απόφαση του δικαστηρίου, θα εξετάσουμε στις 4 Δεκεμβρίου αναλυτικά τις επιλογές που έχουμε. Τώρα, νομίζω ότι εδώ έχω απαντήσει στην κυρία Γιάλα Σέντερ, λέει ο μιλητής, για τι ερωτήσει του κυρίου Σαλαφράγκα. Η κατάσταση με την εκόπωση, το burnout ε, είναι και για μας δύσκολη. Έχουμε 7 burnouts, λέει ο μιλητής. κάτι που προσπαθούμε να προλάβουμε μέσω ευαισθητοποίησης ειδικών καταρτήσεων κτλ. Για, για, τις, για το κόστος των μισθώσεων ε, θα επανέλθω με λεπτομερέστερα στοιχεία αλλά είμαστε σε μια αντίστοιχη κατάσταση με αυτή που εξέφερασε ο συνάδελφος για την ΕΟΚΕ για τους υπολογισμούς Brexit. Ευθυγραμμιζόμαστε και εμείς για τα 24 μέλη που θα προχωρήσουν, με μειώσεις δηλαδή που κονδυλίων που δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα Μπορώ να σας πω ότι το 2017 είχαμε την πρώτη δράση ερωτηματολογίου ικανοποίηση του προσωπικού και σημειώθηκε υψηλό ποσοστό ικανοποίησης που ήταν πάνω από το μέσο όρο των υπολείπων θεσμικών οργάνων. Δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχουν περιοχές στις οποίες πρέπει να βελτιωθούμε και γι' αυτό το λόγο διενεργήσαμε και κάποιες συνεντεύξεις προ-αποχώρησης, αν καταλάβουμε καλά τον ομιλητή. Για τον κύριο Ντεγιόν, Με ευχαριστεί η ερώτησή σα, διότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικοινωνούμε καλύτερα τα πράγματα προς εσά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να το υπογραμμίσω με χοντρό μαρκαδόρο. Τα, ε, οι 180 εκδηλώσεις αυτές στις οποίες αναφερθήκατε ήταν δικές μας εκδηλώσεις. Είναι πολύ σημαντικό προσεγγίσαμε 40.000 πολίτες από μόνοι μας. Και εδώ έχω αποδείξεις. Θα σας δώσω αυτό το έντυπο κύριε Ντεγιόγκ με μεγάλη χαρά για τις εκδηλώσεις που κάναμε και θα το αποστείλουμε και στο Συμβούλιο ζητώντας τους να προσαρτήσουν τα αποτελέσματα στα ε, πορίσματα του Συμβουλίου, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Έχουμε έρθει σε επαφή με τον κύριο Τούσκ σχετικά με το θέμα αυτό και μας ρωτάτε τι μπορούμε να προσφέρουμε στους δυνητικούς επισκέπτες. Εμείς δεν είμαστε πλούσια επιτροπή, δεν έχουμε τέτοιο όμορφο μουσείο που έχετε εσείς, αλλά έχουμε ξεκινήσει εικονικές επισκέψεις, online προγράμματα κατάρτισης για την περιφερειακή πολιτική, για, τα, για ζητήματα δημοκρατίας λοιπά, Τακτικές, τα, τακτικά προγράμματα κατάρτισης κάνουμε και μάλιστα είμαστε το, η το πρώτο θεσμικό όργανο που κάνει κάτι τέτοιο και ετησίως έχουμε 40.000 επισκέπτες, αν ακούσαμε καλά, Επίσης έχουμε συγκεκριμένη ομάδα εργασίας ε, και ε, προετοιμασίας για το Brexit. Έχουμε επισκεφθεί την Ιρλανδία, το θέμα των συνόρων. Βλέπουμε ιδιαίτερη πρόκληση για τις περιφέρειες γιατί τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα σε επίπεδο κράτους μέλους πρέπει να ε, εντείνουμε την προσπάθεια σε περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχουν διάφορα μέσα, έχουμε, έχουμε συγκεκριμένη έκθεση για το θέμα αυτό. Έχουμε κάποιες ομαδοποίηση εδαφικής συνεργασίας. Ο εντατικός διάλογος συνεχίζεται σχετικά με, τον, με το ασύμετρο αντίκτυπο που θα έχει το Brexit επί των περιφερειών και είμαστε σε επαφή και με τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Σα ευχαριστώ. Αν μπορείτε να μου αποστείλετε αυτό το έγγραφο και εμένα, λέει ο Πρόεδρος, ε, πολύ θα μ' άρεσε. Λοιπόν, ο διαμεσολαβητή, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω τα διάφορα ερωτήματα και κάνω μια απόπραντα να Απλά για συγκεκριμένα νούμερα γραπτό η Επιτροπή πρέπει να ζητήσει και όχι μεμονωμένα μέλη. Για το Flexi Time, νέους κανόνες το 2017 ε, με επιτυχία σε ό,τι αφορά την ε, ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής για το προσωπικό μας. Το νέο σύστημα βοήθησε να αυξηθεί και η ευελιξία ε, του γραφείου μας, ε, να διαχειρίζεται απουσίες. Σε ό,τι δεν αφορά τη χρήση του flexi time και της τηλεεργασίας από άνδρες και γυναίκες, κατάσταση ανταγκλά αυτό το οποίο ήδη αναφέρθηκε και χαρακτηρίζει νομίζω αυτή τη στιγμή όλα τα θεσμικά όργανα απέναντι ε, στην αύξηση ενό νέου εργατικού δυναμικού που συνίσταται στο μεγαλύτερο μέρο από γυναίκε. Η χρήση ουσιαστικά είναι η ίδια μεταξύ των δύο φύλων αναλογικά, αλλά σε απόλυτου αριθμού, ε, οι δυνατότητε ε, είναι περισσότερε, άρα τι χρησιμοποιούμε περισσότερο για την τηλεεργασία και το φλεξάμι θα σας δώσω στοιχεία ό,τι αφορά τους συμβασιούχους και τις δυνατότητες σταδιοδρομίες που τους προσφέρονται ο ή φυσικά και επιδιώκει ε, όλο και πιο υψηλά προφίλ. Όχι αυτός ο σκοπός όμως για τη Γιατί ο στόχος είναι να είμαστε πιο γνωστοί στους πολίτες και πιο κοντά στους πολίτες. Άρα έχουμε συμπεριλάβει περισσότερες δραστηριότητες, ε, πιο πολλές ε, έρευνες στρατηγικού είδους και λοιπές ε, στις δραστηριότητές μας με τους περιορισμένους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Όπως είπα, εγώ ξεκίνησα από 1η Σεπτεμβρίου τα καθήκοντά μου ως Γενική Διευθύντρια, ως Γενική Γραμματέας μάλλον, και πάρα πολύ προσεκτικά μελετώ το οργανόγραμμα, τις αναθέσεις, ε, θέσεων, ε, καθηκόντων και φυσικά όπως και η έτσι και εγώ θα σας στέλνω αναλυτικές αναφορές σε περίπτωση που εντοπίσω οποιαδήποτε ε, περίπτωση που χρήζει διόρθωσης. Θα τα θέσω αυτά τα θέματα και είμαι και στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε και σε άλλη ευκαιρία το θέμα αυτό. Στις αποστολές τώρα της Σολαβήτριας. Να ξαναγυρίσω σε ένα θέμα που έρχεται και ξανάρχεται στη συζήτηση. Προσπαθούμε να είμαστε πιο αισθητοί ως ε, για να έρθουν πιο κοντά στους πολίτες όπως είπα. Οπότε, σε σχέση με αυτό σίγουρα η διαμεσολαβήτρια κάνει και αποστολές ε, για να έρθει σε επαφή με τους πολίτες. Μάσκη επιρροής, ε, προσπάθεια επίτευξη πολλαπλασιαστικού αποτελέσματο. Αυτά μπορείτε να τα δείτε όμως πάρα πολύ εύκολα στην ιστοσελίδα μας. Αν θέλετε όμως να σας δώσω και εγώ στοιχεία πιο πολλά για τις αποστολές, ευχαριστώ να το κάνω εφόσον το ζητήσετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επιθεωρητή ε, προστασία προσωπικών δεδομένων, παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ και πολύ σύντομα. Ευχαριστώ καταρχάς για τις ε, ε, γενικέ παρατηρήσεις την κυρία Γιάλα και τον κύριο Σαλαφράνκα. φερθήκατε στην ανάπτυξη του θεσμού μας, του φορέα μας, πολύ σημαντική και λόγω της αύξησης των αναγκών σε προστασία προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστούμε λοιπόν για κάθε υποστήριξη που μας προσφέρετε γιατί χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους. Ε, προσπαθούμε να καταγράψουμε το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης με αυτό που καταγράφεται ή θα καταγραφεί από τους εθνικούς φορείς προστασία προσωπικών δεδομένων. Ξέρουμε ότι θα είναι αρκετό αλλά προσπαθούμε γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι εάν ορίζεται στις αρχές εθνικές ένα συγκεκριμένο ποσοστό στο οποίο υποχρεούνται να προσαρμοστούν, έτσι θα πρέπει να πράξουμε κι εμείς. Ε, πάντως αναφέρατε το νέο διοικητικό Συμβούλιο, Κομιτέ Ευρωπαίου Προτάσεων Τεντάτος, το νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Ε, προχωρούμε με βάση μια οδηγία, δηλαδή εθνική νομοθεσία, εθνική εφαρμογή, εθνικές αρχές, σαν βάση. Και τώρα πέραμε σε έναν κανονισμό, ευρωπαϊκή νομοθεσία δηλαδή, με άμεση εφαρμογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που πρέπει να εγγραφεί στο πλαίσιο μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Προσωπικών Δεδομένων, που όμως δεν ήταν δυνατόν ε, να έχει ήδη συσταθεί. Άρα θεσπίστηκε ένας νέος φορέας, ο οποίος συντονίζει μόνο τις εθνικές αρχές. Αλλά για να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή διάσταση, η γραμματεία της εν λόγω επιτροπής ε, υπήρχε στην EDPS ε, και έτσι στον, στην Ευρωπαϊκή, δηλαδή στον Ευρωπαϊκό Φορέα Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Επιθεωρητή Προσωπικών Δεδομένων και έτσι έχουμε κάνει και οικονομία σε πόρους και σε χρήμα. Στο module που βλέπετε, κύριε Σαλαφράνκα, μιλούμε για το διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν ε, διατεθειμένη να περάσει σε μια συνομιλία με την υπηρεσία μας για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων στους ανθρωπίνους πόρους, αλλά Βλέπουμε μια κάποια αλλαγή τώρα. Μόλις ενημερώθηκα ότι άνοιξε η δυνατότητα για μια συνάντηση την Παρασκευή για να συστήσουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο ε, γίνεται αυτή η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Άρα σε προσεχή συνεδρίαση, συνάντηση θα έχω την ευκαιρία να σας πω περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι έτσι ολοκληρώνουμε το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ τους γενικούς γραμματείς και εισηγητές την εισηγήτρια ε, για τη συμμετοχή τους. Περνώ στο επόμενο θέμα, απαλλαγή για τις ε, υπηρεσίες. Έχω μόνο 15 λεπτά, 10 λεπτά γιατί μετά ανοίγει... Στις 12 ξεκινάμε, άρα έχω 40 λεπτά περίπου, γιατί στις 12 ξεκινάμε την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Παρακαλώ όσοι είναι να αποχωρήσετε, να αποχωρήσετε ησύχως. Okay, I, I'm going to start the in, in 30 seconds. If can you please... Έχουμε, όπως είπα, πολύ λίγη ώρα. Παρακαλώ το ταχύτερο δυνατό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να αποχωρήσουν όσοι να αποχωρήσουν και να εισέλθουν όσοι να εισέλθουν. Παρακαλώ όσοι είναι να αποχωρήσετε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο σημείο που είναι οι απαλλαγίε ε, των κοινών επιχειρήσεων. Έρχομαι την κυρία Γκάλ Πέλτσε από το ελεκτικό συνέδριο. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας, είσαστε και πρώην μέλος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι με μεγάλη χαρά βρίσκομαι και πάλι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ξαναβλέπω, βλέπω πολλά γνώριμα πρόσωπα για την έκθεσή μας ε, επί των ε, κοινών επιχειρήσεων για το 2017. Όπως κάθε χρόνο ε, εκδώσαμε έκθεση σχετικά με την αξιοπιστία και την ακρίβεια των μεγεθών και των σχετικών συναλλαγών. Μιλούμε για συμπράξεις ε, δημοσίου ιδιωτικού φορέα στα κράτη-μέλη που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για, συγκε... για συγκεκριμένες πτυχές ε, της ε, υλοποίησης ευρωπαϊκής πολιτικής. Το 2017 είχαμε 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικό προϋπολογισμό σε σχέση με 2,8 αν ακούσαμε καλά το 16 και σύμφωνα προς τον προϋπολογισμό του προϋπολογισμού είχαμε ανεξάρτητες, ε, ε, ανεξάρτητους εξωτερικούς ελέγχους για όλους, όλες τις κοινέ επιχειρήσεις έχουμε λάβει επαρκείς εγγυήσεις ε, για την δουλειά που έκαναν αυτοί οι εξωτερικοί ανεξάρτητοι ελεγκτές. Σχετικά λοιπόν με την αξιοπιστία των λογαριασμών. Το 17 σχετικά με τα αποτελέσματα και τις οικονομικές ε, θέσεις και τις ε, ροές έχουμε μια καθαρή θέση και για τις οκτώ κοινέ επιχειρήσεις για τις συναλλαγές νομικές ή μάλλον νομότυπες ε, και κανονικές για όλα τα GUs εκτός από την Excel για λόγω της μη εναρμονισμένης ε, μεθοδολογίας ε, των ε, εθνικών αρχών χρηματοδότησης. Αυτό βέβαια το θέμα απλώς αν... αναφέρεται σε πληρωμές FP7, λέει η ομιλήτρια. FP7 αλλά είμαστε σε, σε φάση σταδιακής απόσυρση του FP7 και κανονικά θα πρέπει να εκλείψει για τα επόμενα χρόνια. Όπως και το 16 για το Fusion for Energy σημειώνουμε τα θετικά βήματα που έχουν αναλυφθεί για να βελτιωθεί η διοίκηση και ο έλεγχος, αλλά θέλαμε να συστήσουμε την ε, ε, προσοχή τους για τον κίνδυνο περαιτέρω αύξησης ε, κόστους. Πέραν αυτού και όπως γνωρίζετε το 2017 ολοκληρώσαμε τις τελικές αξιολογήσεις ε, για τις κοινέ επιχειρήσεις υπό το FP7 και τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις για τον ορίζοντα 2020. Συνολικά ήταν θετική θετικός ο έλεγχος, είχαμε κάποιες συστάσεις και κάθε κοινή επιχείρηση προετοίμασε σχέδιο δράσης ε, που ξεκίνησε να, ελέ... να υλοποιεί το 2018. Στους ελέγχους το 2018 θα παρακολουθήσουμε από πλευρά ελεγκτικού συνεδρίου την υλοποίηση αυτών των σχεδίων δράσεων. Για τον ορίζοντα 2020 και το FP7 επέτυχαν ένα συνολικό ε, ποσοστό υλοποίηση 82% για το FP7 και 23% για τον ορίζοντα 2020. Και για να συνοψίσω, η έλεγχοι του 2017 επιβεβαιώνουν τα θετικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών. Χαιρετίζουμε το γεγονό ότι οι κοινέ επιχειρήσει έλαβαν ε, διορθωτικά μέτρα σε σχέση με, με τα προηγούμενα έτη ε, στοιχεία που χρήζουν τις προσοχής της διοίκησης είναι δημοσιονομικά και χρηματοπιστωτικής διαχείρισης εσωτερικών ελέγχων και εισφορών. Συμπερασματικά για το 2017 έχουμε 8 καθαρές εκθέσεις για την αξιοπιστία των λογαριασμών, μία ε, σχετικά με την Excel για την νομιμότητα και τακτικότητα των συναλλαγών και μία έμφαση ε, για την ε, Fusion for Energy. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Για να κερδίσουμε ίσως λίγο χρώμο, αντί να πάμε στις κοινέ επιχειρήσεις, θα πάμε στους ε, εισηγητές. Παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις ε, που νομίζω ότι είναι απαραίτητες ε, και μετά έχω και τέσσερις ερωτήσεις Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, γιατί βελτιώσατε την έκθεση μας ότι αφορά τις κοινές επιχειρήσεις που δίνει πολύ συνοπτικές καλές πληροφορίες. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τις κοινές επιχειρήσεις. Κάνουν πολύ καλή δουλειά, συνεισφέρουν στο ερευνητικό θεματολόγιο της Ένωσης. Όμως ε, θέλω πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είχαμε αυτή τη δέσμη δεδομένων στην ενδιάμεση αξιολόγηση των ε, κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020. Ήταν εξαιρετικά τα δεδομένα και σε αυτά έπρεπε άλλωστε και να βασιστούμε. Για την αξιολόγηση τώρα της προστέμενης αξίας. Στον κατάλογο μου πάντα έχω την έρευνα, την καινοτομία και την παιδεία. Ορίζον 2020 και τα πριν και μετά προγράμματα δείχνουν ότι δεν αρκεί ε, να γίνει μια καλή χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων, αλλά το ταλέντο, η κινητικότητα, η γνώση μπορούν να ενισχύσουν την Ένωση απέναντι στους παγκόσμιους ε, εταίρους μας. Οι κοινές επιχειρήσεις ε, συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη, την δημιουργία θέσεων Εργασίες και σας ευχαριστώ κοινές εκμεταλλεύσεις. Ό,τι αφορά ιδίω ε, το ορίζον 2020 έχουμε αυτές τις κοινοπραξίες. Είναι σημαντικό γιατί έτσι μπορούν να κινητοποιήσουν και να συνενώσουν ένα κατακαιρματισμένο τοπίο ε, και κλάδους. Και κάποιοι εμπλεκόμενοι που κανείς δεν θα φανταζόταν ίσως ότι ε, μπορεί να συνεργαστούν, μπορούν να συνεργαστούν τελικά μεταξύ τους. Και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα και πρέπει να το αντιληφθούμε. Χαίρομαι λοιπόν που οι κοινέ επιχειρήσει ε, κινητοποιούνται όχι μόνο για ε, του ιδιωτικού και δημόσιου πόρου που θα κληθούν να διαχειριστούν, αλλά και γιατί γίνονται πρωταγωνιστέ, ηγέτε. Όπω είπε και το Ελληνικό Συνέδριο, όμω ε, παρά τις, τα επιτεύγματα, ζητείται συμμετοχή μεγαλύτερου φάσματος εμπλεκομένων φορέων στις κυβερνητικές δομές, δομές διακυβέρνηση δηλαδή, ή στις κοινοπαραξίες που συμμετέχουν σε έργα. Ε, έχουμε λοιπόν στους εκπροσώπους των κοινών επιχειρήσεων που έχουμε εδώ παρόντες. Αυτή η αύξηση της συμμετοχή κρατών μελών, άλλων φορέων, ε, της βιομηχανίας, ΜΜΕ και άλλων. Είναι κάτι εφικτό, εν γέννη. Και η περαιτέρω διαδικτύωση με κοινοπραξίες και κοινέ επιχειρήσεις μπορεί να αυξήσει την βιωσιμότητα και την προσθέμενη αξία των έργων αυτό λοιπόν το αίτημα των εμπειρογνωμόνων που ζητούν μεγαλύτερη συμμετοχή, πώ το βλέπετε, σε ό,τι αφορά τώρα τι επιδόσει ε, και την κοστομηνία. Ξέρετε ότι ε, μου είναι ιδιαίτερα προσφύλλα αυτά τα θέματα. Μιλάω για επιδόσει και ευρωπαϊκή προσταμινή αξία. Δεν ε, εστιάζομαι σε αυτό το πολυματικό περιθώριο σφάλματο ή στι μικρέ αδυναμίε και ανεπάρκειε σε ό,τι αφορά και τι δημόσιες προμηθείες, σε ό,τι δεν αφορά τους δείκτες. Αντίθετα από το 7ο πρόγραμμα, πλαίσιο στο Horizon 2020 θέλω να δω τις τρεις δέσμες δικτών για να βελτιωθεί ο αντίκτυπος, να γίνει κατανοητή η στρατηγική πρόκληση από την πλευρά όλων των φορέων και για να αιτιολογηθεί και υποστήριξη προς τα μέσα των κοινών αυτών επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τη μέτρηση της πλειοψηφίας των ε, δικτών των βασικών δικτών επιδόσεων. Ε, ξέρω ότι δεν είναι εφικτό τώρα ε, να τους μετρήσετε από κοινό, αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει στο μέλλον για να μπορούμε να τους καταλάβουμε καλύτερα. Άρα ελπίζω να μας δώσετε πραγματικά νούμερα, απτά αποτελέσματα στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά την διάμεση αξιολόγηση. Ε, οι συντονιστές είπαν ότι το 34% μόνο των έργων πέτυχαν πλήρω του στόχου του και αυτό με ανησυχεί. και λέει επίσης ότι κάποια ε, πέτυχαν και κάποιους στόχους που δεν ήταν αναμενόμενοι και είχαν ε, κάτι πολύ, ε, αυτό ήταν κάτι πολύ θετικό και το 49 των έργων, ούτε το μισό, με μικρές αποκλήσεις πέτυχαν τους στόχους τους λίγο πολύ. Και τις δίκαινες επιχειρήσεις και την Κομισιόν. Θέλω να ρωτήσω, ποια είναι τα βασικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν την επιτρέψη όλων των στόχων από τις ε, κοινέ επιχειρήσεις, από τα έργα. Θα βοηθούσε το να υπάρχει αυτός ο, αυτό το κοινό πλαίσιο με τους βασικούς δείκτες. Θα σας πω τι μπορούμε να κάνουμε. Και όπως λέει και το ελεκτικό στην έκθεσή του, στα τέλη του 17, κοινή διαχείριση επιχορηγήσεων και εργαλεία παρακολούθηση για το 2020 δεν είχαν οδηγήσει σε μεγαλύτερες σε είδος συνεισφορές. Και μιλάμε για τέσσερις ε, επιχειρήσεις. Αυτό το εργαλείο το οποίο αναφέρεται πότε θα είναι έτοιμο και τελευταίο ενημερώθηκα ότι ο πρόσφατο κανονισμό δεν είναι και τόσο ευνοϊκός απέναντι στην πιο στενή συνεργασία μεταξύ των κοινών επιχειρήσεων. Κάτι που θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την προσθέμενη αξία με συνέργειες, με κοινή χρήση πόρων και γνώσης ανταλλαγή διδαγμάτων. Δεν ξέρω, κοινέ προκήρυξεις διαγωνισμών για παράδειγμα ή ε, καινοτομία που θα την ε, μοιράζονται κάποιες κοινέ επιχειρήσεις. Τελευταία ερώτηση. Όλοι οι φορείς τι έχουν να πούν για αυτό που είπα και γιατί δεν το θέλουμε. Ποιο είναι το εμπόδιο, γιατί δεν θέλουμε μεγαλύτερη συνεργασία. Σταματώ εδώ για τα γενικά. Και θα ακούσω ε, με τα χαρά της παρουσιάσει ερωτήσει σα. Straight to Ας πέρασουμε στο σκιώδης αμέσως, ο κύριος Βετσόφσκι. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τη Μαρτίνα Κλαμπάγιοβα, το Ευρωπαϊκό Λεκτικό Συνέδριο και τον πολύ καλή συνάδελφο που είναι εδώ, που κάθε φορά μα προσφέρει εξαιρετικά και χαίρομαι που έχουμε εδώ τόσο καλούς εκπροσώπους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και περνάω αμέσως στα τσεχικά για να πω ότι ήθελα να παρακολουθήσω την υπόθεση, όπως είπε και η συγγήτρια. Μπορούμε να βελτιώσουμε την κοινή δράση, την κοινή διαχείριση. και σε σχέση με την... Ε, με την ε, διαχείριση λοιπόν πρέπει να απλουστεύσουμε το έργο των κοινών επιχειρήσεων χωρίς όμως περιορισμούς ε, ή συμβιβασμούς στην αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια. Πρέπει να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα χρηματοδότησης σε πολλαπλά επίπεδα. Χρειαζόμαστε απλοποίηση στα οικονομικά. Καθώς έχουμε τρία επίπεδα στο ECSL, το τρικοματικό, το, σε, τρία επίπεδα, δηλαδή το ορίζον, το εθνικό και το επίπεδο συμμετοχής της, ε, του κλάδου. Σε αυτό μπορούμε να έχουμε μία απλοποίηση για να έχουμε και καλύτερη ε, ορατότητα στις κοινέ επιχειρήσεις. Και καλό, απευθύνω έκκληση προς όλες τις κοινέ επιχειρήσεις. Ανοίξτε τις... Ε, ε, στραφείτε προς το κοινό, προσπαθήστε να πείσετε, να πουλήσετε ούτως οπίν τις επιχειρήσεις σας, τα έργα σας στο κοινό, στον πολίτη. Και πάντα εδώ έχουμε την αρχή της επικουρικότητας, δηλαδή ότι καλύτερα γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντί για το εθνικό, θα γίνεται σε ευρωπαϊκό. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Η Ευρώπη έχει πολύ καλές δυνατότητε για ανάπτυξη δραστηριοτήτων με βάση τι κοινέ επιχειρήσει, στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωση, είναι να ηγηθούμε στην έρευνα και την καινοτομία. Πρέπει να αναπτύξουμε και, στον, και τον κλάδο των κοινωνικών συνεπειών των ε, ε, των, ε, των κοινών επιχειρήσεων. Ο κύριο Πός. Και ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Προπολογισμό κοινές επιχειρήσεις και έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτούμε καλύτερα τα στοιχεία που παρουσιάζουν βελτίωση αλλά και τα προβλήματα. Ο Ορίζον 2020 είχε πλήρη εφαρμογή. Έχω βάλει άλλα ακουστικά. Η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη. Προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε τα, τα καταλληλότερα δυνατά αποτελέσματα. 23% κατά μέσο όρο στα προγράμματα. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό. Ε, αν συνεχιστεί και το 18 βεβαιώνεται η θετική τάση. Σχόλια και ερωτήσεις από πλευράς μου. Το ελεγκτικό συνέδριο λέει ότι το τέλος του 2000, στο τέλος του 2017 δεν είχε ολοκληρωθεί η ανάπτυξη ορισμένου τομεί όπως παρακολούθηση της ε, διαχείριση των ποσών και κυρίως σε υλικό επίπεδο. Ε, μπορείτε να μας δώσετε πιο πολλές λεπτομέρειες. Τι συνέπειες μπορεί να είχε αυτό στην ε, διαδικασία διαχείρισης των κοινών επιχειρήσεων και έχουν αναλυφθεί διορθωτικές κινήσεις. Επίσης είχε υπογραμμίσει το ελεγκτικό συνέδριο της συνέπειας του Brexit και της αποχώρησης από την Ευρατόμ, της σύνδεξης για την Ευρώπη. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις εδώ. Στο μέλλον του Ηνωμένου Βασίλειου θα συμμετέχει στον προπολογισμό θα συμβάλλει σε αυτές τις κοινέ επιχειρήσεις και με ποια μορφή. Στο ίτερ, επί παραδείγματι, τι είδους συνέπειες θα έχει για το μέλλον. Και επίσης έχουμε ένα χαμηλό ποσοστό συμμετοχής Υπήρχε μία πρόταση νομίζω που ήθελε η κοινή επιχείρηση κάποια κονδύλια να τα κρατήσει για ορισμένα έργα και αποφάσισε να μην απορροφήσει όλα τα ποσά, 17% μόνο, που είναι πάρα πολύ χαμηλό. Ε, αλλαγή του κανονισμού που επιτρέπει εξωτερική χρηματοδότηση προχώρησε γρηγορότερα για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι για τις προκηρύξεις ε, την Άνοιξη. Έγινε αυτό. Γιατί είχαμε κάποιες ε, αποκλήσεις. Ελπίζω μόνο να, έχουν βελτιωθεί, να έχει βελτιωθεί η εικόνα. Εν τω μεταξύ, καλώς, ευχαριστώ και τώρα περνούμε στις απαντήσεις από τις ίδιες τις κοινέ επιχειρήσεις, στις ερωτήσεις των συναδέλφων μας. Σφέμα. Το σύνδεξη για την Ευρώπη, F4E, κύριε Σφέμα. Πέντε λεπτά. Χαίρετε Σφέμερ και είμαι ο Διευθυντής του Fusion for Energy. Συνήθως η φωνή μου είναι πιο ευχάριστη, με συγχωρείτε όμως είμαι βραχνιασμένο σήμερα. Νομίζω ότι με διευκολύνει κιόλα ε, το ότι μου περιορίζεται το χρόνο στα πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ τον Αντιπρόεδρο κύριο Βόν και ιδιαίτερα την κυρία Λαβάρσοβα, Αντιπρόεδρο και εισηγήτρια, για την ευκαιρία να σας μιλήσω σήμερα εδώ και να σα παρουσιάσω τι θέσει μα. Τι ήθελα να πω λοιπόν ε, Θα να εκφράσω την ε, ικανοποίησή μου για την ε, θετική ανταπόκριση του ελεγκτικού συνεδρίου στις εκθέσεις μας. Ε, με χαρά να απαντήσουμε και στις ερωτήσεις που έχουν διατυπωθεί ευθύς αμέσως λαμβανομένων υπόψη ε, των περίπλοκων στοιχείων ε, του έργου μας. Ε, καλωσορίζουμε την χωρίς επιφυλάξεις έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν θα σας διαβάσω όλο το κείμενο βέβαια. Παρατηρήσεις του συνεδρίου. Πιο λεπτό μερός, καθώς είναι αρκετά περίπλοκο και ρυψοκίνδυνο το έργο. Διαδικαστικά έχουμε ε, ιστορικούς ελέγχους, τους ενισχύουμε στους τομείς του οικονομικού σχεδιασμού και της επιλογής και πρόσληψης προσωπικού με βάση και τις ε, εκθέσεις του συνεδρίου με βάση και τις βελτιώσεις που έχουμε στην βελτίωση, στην ε, εξοικονόμηση πόρων το 2016, συνεχίζουμε. Έργα όπως το ITER συνεχίζονται με παλιθεύσεις και προκαταβολική αξιολόγηση κινδύνου συνεχίζουμε στις προηγούμενες δράσεις που έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραδείγμα τη συμφωνία με το ΙΤΕΡ για τη βελτίωση των οροσίμων, αλλά και για την ε, καταγραφή της επιπλέον αξίας, της επιπλέον εξασφαλιστής αξίας, αλλά και οικονομική αξιολόγηση του ΙΤΕΡ, για την οποία θα σας δείξω κάποιες διαφάνειες που οι διερμηνείς δεν μπορούν να δούνε. και συνεχίζουμε τις διαδικασίες με βάση τον οικονομικό κανονισμό. Θα ήθελα κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, κάποια σημεία ιδιαίτερα να τονίσω. Έχουμε ακολουθήσει τις συστάσεις ε, για τις δράσεις ε, του ελέγχου σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Συστηματικά ε, επαληθεύουμε εσωτερικά και ολοκληρώνουμε τα πρώτα πέντε. Έχουμε ενισχυμένα συστήματα και χρησιμοποιούμε και το KPI που είναι διαθέσιμο. Έχει βελτιωθεί το πρόγραμμα με σημαντικό αριθμό προσωπικού διαχείρισης και η έρευνα προσωπικού σημειώνει πρόοδο ελαφρά γιατί βελτιώνεται ο έλεγχος και η λειτουργία στη διοίκηση. Οι αλλαγές δεν γίνονται κατανοητές από το προσωπικό μας. Update on the status of the e project, which you can see evolving here on the picture while I'm talking. Εν τω μεταξύ εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε τις διαφάνειες στην οθόνη όσο όμιλο και σας καλώ τώρα να δείτε την φωτογραφία από το Ίτερ με κατασκευή, με ένα εργοτάξιο εντυπωσιακό. Η κυρία Μαλόβα ήρθε και μας επισκέφθηκε η ίδια. Φαντάζομαι ότι θα έχει και δύο λόγια να πει για τις εντυπώσεις που συνέλεξε. 2.000 εργαζόμενοι με 2,5 βάρδιες τη νύχτα παραδίδεται το υλικό. Και ο εξοπλισμός από τους βιομηχανικούς εταίρους καταφθάνει διαρκώς. Yeah. So um, I still remember when I talked first to Mrs. Dressler and she said την κυρία Γκρέσλε. Μας είπε, α, είναι ελεκτικό συνέδριο εδώ, είναι έλεγχος προπολογισμού εδώ, δείξτε μα τι έχετε κλείσει ω μέργο. Να λοιπόν, τελειώσαμε την πρώτη πηγή ακτίνας ε, εγκαταστάσει. ε, Σας περιμένουμε να τις δείτε. Είναι, νομίζω αυτό ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα που αποδεικνύουν ότι η δουλειά γίνεται. και έχουμε τη δυνατότητα δοκιμής της ε, ε, θέρμανσης της ουδέτερης ακτίνας του, B, του Ίντερ. Και κοιτώ τώρα τις, ε, τον αντίκτυπο στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε περάσει τα 6 λεπτά, μας έχουν μείνει 11 για να κλείσουμε. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν θέλετε να στερήσετε από τους άλλους συναδέλφους σας ε, το χρονομιλίες. Καλά, να τελειώσω πιο γρήγορα τότε, Πρόεδρε. 40.000 ε, χρόνια έχουν παραχθεί, έτσι. το βλέπετε άλλωστε, αύξηση του όγκου ε, που είναι ωφέλιμος και για, την, ε, για τον κλάδο και κλείνω πολύ στόμα με τα συμπεράσματα ότι καλωσορίζουμε την γνώμη του συνεδρίου, τα αποτελέσματα μας είναι θετικά, έχουμε περάσει πλέον σε ένα σημείο που είναι βέβαιη η λειτουργία και η αποδοτικότητα, δεν υπάρχει επιστροφή, προϋπολογισμός μέσα στα πλαίσια του, Πουλου, του 2020 και σας ευχαριστώ πολύ αν υπάρχει η δυνατότητα θα ήθελα να φερθώ στις ερωτήσεις. Συγκεκριμένα για το Brexit, ξέρετε ότι Έχουμε χρηματοδότηση από τη συνθήκη της Euratom με συνδεδεμένη χώρα την Ελβετία και μηνύματα από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι στιγμή πώ θα ενδιαφερόταν για αντίστοιχη μορφή συνεργασία σύνδεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει την εντολή από το Συμβουλίο για την ανάληψη των διαπραγματεύσεων. Όπω είπε ο κ. νωρίτερα είναι μια εξέλιξη που αναμένεται στο μέλλον, άρα δεν μπορούμε να την προβλέψουμε. Πάντω, αν όλα πάνε καλά, μέσα σε δύο χρόνια θα έχουμε πιστεύω τη δυνατότητα διασύνδεσης και με τη μεταβατική περίοδο, έτσι ώστε να προχωρήσει η μετάβαση χωρίς κλειδονισμούς. Η βέλτιστη εκδοχή είναι αυτή βεβαίω πιο αισιόδοξη. Πιστεύουμε όμως ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Βέβαια σε περίπτωση hard Brexit, δηλαδή Brexit χωρίς συμφωνία, δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει, να προκύψει Η απόφαση ε, εναπόκειται στους αρμόδιους για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων και όχι σε εμά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να περάσουμε στο Excel. Ο κύριος Κομπανία, αν ακούσαμε καλά, είναι ο Γενικός Διευθυντής. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα, αλλά ξεκινώντας από το εξής. Εχθές το βράδυ, λίγο πριν τις 9, κοιτούσα στο iPad ε, για την ε, προσαρίωση του σκάφους που στείλαμε, που έστειλε η NASA, και αναζητούσα στη Wikipedia όλα, όλο τον εξοπλισμό σε αυτό το 50 κιλών σκάφος όλα αυτά ήταν φτιαγμένα στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πολύ ενδιαφέρον πως το Made in Europe είναι πλέον διαθέσιμο στον Άρη. Όλη αυτή η τεχνολογία είναι, περνάει από ένα πολύ περίπλοκο μείγμα εξοπλισμού δεν ε, φτιάχνουμε λειτουργικά προγράμματα και chips επειδή μας αρέσει, ε, αλλά επειδή επιτρέπει σε άλλους να κάνουν τη δική τους δουλειά, για παράδειγμα, να πηγαίνουν στον Άρη. Σχετικά με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων, έχω αυτό που κρατάω στο χέρι μου, που είναι μια ευφυής ένα ευφυή καθετήρας, ο οποίος μέσω μια συσκευή θέρμανση μπορεί να προχωρήσει σε μικρές διορθώσεις προς τον μη που είναι η καρδιά, ώστε να αυξάνει το προσδόκιμο ζωής ε, διορθώνοντας ε, κάποιες ε, δυσλειτουργίες της καρδιάς. Επίσης έχουμε μια σειρά από ενδιαφέροντα έργα στην Αυστρία ανακοινώθηκε 1,5 δισεκατομμύριο επένδυση για εργαστήριο ε, μικροτσίπ στα Power Electronics που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο αλλά κυρίως ε, επιτρέπει την κυκλοφορία των ηλεκτρονικών οχημάτων ώστε να μετακινηθούμε από το ρηκτά καύσιμα στα ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρική ενέργεια σε πιο αποδοτικές ενεργειακές ε, εφαρμογές. Αυτό δείχνει τη δραστηριότητα μέσω Excel και τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Για το υπόλοιπο των δραστηριοτήτων μας να αναφερθώ στο συνέδριο στο ημικύκλιο σήμερα το απόγευμα για την έρευνα και την καινοτομία που θα δείτε όχι μόνο τον καθετήρα αλλά θα έχετε και τον κύριο Πικάρ που θα εξηγήσει πώς θα μπορούσε να πετάξει στο Solar Impulse γύρω από τον πλανήτη ε, χρησιμοποιώντας ε, την ηλιακή ενέργεια. Με την πίεση του χρόνου να σας πω απλώς ένα-δυο πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε εν είδη βελτιώσεων μας ε, μίλησαν για τα πολλαπλά επίπεδα των επιχειρήσεων. Έχουμε πράγματι τρία επίπεδα συγχρηματοδότησης, το οποίο αρχικά το είχαμε ε, συστήσει σε ένα σύστημα τριών επιπέδων εκθέσεων σχετικά με τους, ε, τα οικονομικά στοιχεία που λαμβάνουν και τους λογαριασμούς που λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη. Ε, σχετικά με την υποβολή εκθέσεων δημοσιονομικών έχουμε από τα κράτη-μέλη και από την Κομισιόν Ιδανικά θα έπρεπε να έχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων για την υποβολή οικονομικών εκθέσεων, το οποίο πλαίσιο έχει ήδη βελτιωθεί από τα κράτη-μέλη, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε κοινού κανόνες ε, ε, για την αξιολόγηση των ε, χρηματοδοτικών εισφορών των συμμετεχόντων, κρατών μιλών δηλαδή και Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντω αυτό το τριμερέ είναι ένα μοναδικό σύστημα γιατί μπορέσαμε να συνεργαστούμε για να φτάσουμε σε μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική ηλεκτρονικού εξοπλισμού που τη μοιραζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη και τους, ε, τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επίσης, συνεργαζόμαστε πολύ στενά για να αναπτύξουμε ένα οικοσύστημα αν δείτε άλλα μέρη του κόσμου, κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο όπως η Κίνα ή οι Ηνωμένε Πολιτείε. Σχετικά τώρα με την υποβολή έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου ε, που δεν έχει καμία σχέση με τα έσοδα, είναι ένα θέμα υπό το FP7 όπου έχουμε καταποκοπήν ποσοστό ε, σχετικά με το κόστος που αναγνωρίζουν το κράτη-μέλη διότι λόγω της περιορισμένης αρμοδιότητας ε, δεν μπορεί να τοποθετηθεί διαφορετικά το ελεγκτικό συνέδριο. Ζητούμε λοιπόν από καθένα από τα κράτη-μέλη μια ε, δήλωση διασφάλισης ποιότητας ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλα, όλες οι δαπάνες των κρατών μελών έχουν ε, λάβει χώρα με τον σωστό τρόπο. Σε, ευχαριστώ πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη για τα λίγα δευτερόλεπτα που υπερεύει το χρόνο. Ευχαριστώ. Σίζα Τώρα ο κύριος Φρέσνο. Γεια σας και ευχαριστώ. Ναι, εδώ είμαι πίσω εκεί. Πρώτα απ' όλα ε, είναι δύσκολο μέσα σε πέντε λεπτά. Ο εκτελεστικός μας διευθυντής ε, Γκυγέρμη δεν μπορούσε να είναι εδώ. Εγώ λέγομαι Χωσέ Αντώνιο Κάλβο. Uh, Administration Affairs at, uh, the to try και θα προσπαθήσω να σας δώσω όποια εξήγηση χρειαστείτε. Και βέβαια, αν χρειαστείτε και άλλες πληροφορίες ή το εκτελεστικό διευθυντή, είτε εγώ προσωπικά, θα εκπονήσουμε οποιοδήποτε έγγραφο, οποιαδήποτε εξήγηση θέλετε, θα σας τη στείλουμε γραπτό. Είμαστε στη διάθεσή σας. Yes, ε, 2017 has Το 2017 ήταν ε, κάπως... Ε, ιδιαίτερη χρονιά υπό την έννοια ότι είχαμε το διοικητικό κλείσιμο του ΣΥΖΑΡΕΝΑ, του πρώτου δηλαδή προγράμματος ε, που είχαν ε, χρηματοδοτήσει τα ευρωπαϊκά δίκτυα και το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και φτάσαμε πλέον ε, σε ρυθμό κρουαζιέρας για το ορίζον 2020, με κονδύλια δηλαδή το ορίζοντα 2020. αυτή την έννοια βεβαίως και λάβαμε την έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου. Είδαμε ότι ήταν μια θετική άποψη, καθαρή, καλό αυτό. Φυσικά όλα τα σχόλια και όλες τις παρατηρήσεις τα πήραν πολύ σοβαρά υπόψη μας. Είναι βοήθεια για μας τέτοιες εκθέσεις για να βελτιώσουμε τη χρηματοοικονομική μας διαχείριση, αλλά και από άλλες πτυχές. Όσον αφορά τη στελέχωση, για παράδειγμα, είναι χρήσιμες οι συμβουλές του ελεκτικού. Έρχομαι στα συγκεκριμένα ερωτήματα. Τι έγινε με την εφαρμογή του προπολογισμού το 2017, αυτό ήταν το ερώτημα. Από ό,τι καταλαβαίνω αυτό έχει να κάνει με τον προπολογισμό του Σιζαρένα και είναι σαφή η εξήγηση. Ήταν το τέλος του προγράμματο ε, του Σιζαρένα. Ξέραμε ότι είναι το τελευταίο έτος εφαρμογή ε, του προπολογισμού διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών ε, και 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Ε, τέλειωνε η χρηματοδότηση σιγά σιγά, οπότε έπρεπε να λάβουμε υπόψη οποιοδήποτε ενδεχόμενο να δούμε τι πληρωμές έπρεπε να γίνουν το 17 ή το 18 να αποφύγουμε να μην έχουμε επαρκή χρηματοδότηση για να εξοφλήσουμε τις πληρωμές. Τι έγινε όμως, ε, Μέχρι να ζητήσουμε από την Κομισιόν την τελική, την οριστική πληρωμή, δεν είχαμε τα αποτελέσματα από τις εκθέσεις οικονομικής κατάστασης των μελών μας. Δηλαδή δεν ξέραμε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα συνολικά για το ΣΕΖΑΡΕΝΑ. Αν θα έπρεπε να υπάρξει ανάκτηση ποσών ή καταβολή επιπλέον ποσών λόγω της προχρηματοδότησης και της εκαθάρισης της σχετικής ή από τις οικονομικές εκθέσεις τέλος πάντων. Η στρατηγική θέση είναι να είναι κανείς συντηρητικός στις εκτιμήσεις του για τις αξιώσεις ε, κόστους για τα τέλη του 17 και τις αρχές του 18. Αυτή ήταν η προσέγγιση που ακολουθήσαμε. Να δούμε ποια θα ήταν τα ανώτατα επίπεδα πληρωμών, αν από τις οικονομικές εκθέσεις και τους ελέγχους το 2017 ήταν θετικό ε, το υπόλοιπο, έπρεπε να πληρώσουμε δηλαδή τους δικαιούχους ή αν είχαμε κάποια τιμολόγια που μπορούσαν να έρθουν τελευταία στιγμή και δεν τα περιμέναμε. Και επίσης έπρεπε να δούμε τι θα γίνει με την ανάγκη να επιστρέψουμε χρήματα στα κράτη-μέλη που έδωσαν πιθανόν ε, παραπάνω χρήματα. Τα οποία αυτά τα χρήματα ουσιαστικά τα, τα φυλάξουμε εμείς ε, μέχρι το τέλος του προγράμματος, όπως προβλέπει η νομική πράξη. Τα υπολογίσαμε όλα αυτά και έτσι καταλήξαμε στο ποσό που ζητήσαμε από την Κομισιόν. Τελικά, είδαμε ότι ναι, πράγματι ήταν χαμηλή η εκτέλεση του απολογισμού, το είπε και η συγγήτρια. Αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα ουσιαστικά, γιατί εξακολουθούμε να εξοφλούμε τα τελευταία τιμολόγια αυτή τη στιγμή. Άρα του χρόνου θα κάνουμε την τελική καταμέτρηση για το Σέζαρένα και ό,τι έχει απομείνει θα επιστραφεί στην Ένωση. Δεν θα έχει μείνει τίποτα δηλαδή στο τέλος. Τα στοιχεία αφορούν το 17 βέβαια. Γιατί για το ΣΥΖΑΡ ένα συνολικά πρέπει να σας πω το ποσοστό εκτέλεση του προπολογισμού προσεγγίζει το 90% για τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που κάποιες φορές σημαίνει ότι κάποια έργα δεν λειτουργούν και τα κλείνουμε. Είναι υψηλό το ποσοστό αυτό και είμαστε υπερήφανοι για το επίπεδο αυτό εκτέλεσης. Πάντως, όπως και αν έχει, είμαστε στη διάθεσή σας αν θέλετε και άλλες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Έχει περάσει 12, αλλά επειδή η συγκήτρια είχε θέσει ερωτήσει και προ την Κομισιόν και έχουμε εδώ εκπροσώπου τη Κομισιόν. Θα σα παρακαλέσω με ένα-δύο λεπτά να απαντήσουν ε, στι ερωτήσει τη Σύγητρια. Λιμπενέ. Ευχαριστώ. Η πρώτη ερώτηση Σύγητρια αφορούσε κάποια έργα που είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα, πάνω από το 5%. Και αυτό έχει να κάνει με δύο πράγματα. Ο πρώτος λόγος είναι αύξηση της φιλοδοξίας των έργων στη φάση της κατάθεσης πρότασης. Κάθε διαγωνισμό σε πραγματικά ε, συνιστά μεγαλύτερη πρόκληση και οι στόχοι είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτυγχάνονται. Κατά δεύτερος λόγος, η παρακολούθηση αυτών των έργων στη φάση της υλοποίησης είναι πιο αυστηρή και στενή η παρακολούθηση αυτή. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια τάση αυτή και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να την επιβραδύνουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση εδώ. Στην φάση της αξιολόγησης θα πρέπει να κάνουμε τα δέοντα. και για το σχέδιο δράσης. Να είναι αναλογικό των φιλοδοξιών. Να είναι και ρεαλιστικό όμω ταυτόχρονα, να μπορεί να επιτευχθεί. Θα δώσουμε λοιπόν στη βάση τη αξιολόγηση μεγαλύτερη έμφαση στην αναλογικότητα μεταξύ φιλοδοξία του έργου και πόρων που διατίθενται για την επιτευχή τους. Ένα άλλο ερώτημα είχε να κάνει με τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων κοινών επιχειρήσεων. Με το Excel παρακολουθούμε τα πράγματα και από την Γαμματικά Υπάρχει μια πρωτοβουλία από την κοινότητα καινοτόμων φαρμάκων, για παράδειγμα. Και αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε το software και το hardware που θα μας επιτρέψει να κάνουμε τις δοκιμές που είναι απαραίτητες και τα πειράματα σε ιατρική πλατφόρμα θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και συνεχίζουμε τις ε, επαφές ελπίζοντας ότι θα έχουμε ο πρόεδρος ο πρόεδρος απαντήσεις απαντήσεις μόνο τελειώσαμε Um, good morning. Well, it's not good morning anymore. Good afternoon. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ. Με βάση τόσο υπόθηκαν ήδη σήμερα για το Σέζαρ, ενώ όλο πιστεύω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ικανοποιημένη από την εφαρμογή κατά 90 ή και περισσότερο του Σέζαρ σε ένα έργο, ε, στο Brexit Εφόσον υπάρξει συμφωνία, πάντα εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου για την ε, αεροπορία, για την αεροπλοεία. Αυτό είναι μια πρώτη προϋπόθεση για το ΣΕΖΑΡ. Βεβαίω, δεύτερη προϋπόθεση είναι να παραμείνει συνδεμένο στο Horizon 2020 και μετά το Horizon ε, Ευρώπη, του Ηνωμένο Βασιλείου, δηλαδή να συνεχίσει να συμβάλλει στον προϋπολογισμό για τα προγράμματα της Ένωσης. Εφόσον συμβεί αυτό, θα μπορούν και να είναι επιλέξιμε οι αντίστοιχε υπηρεσίε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δύο είναι προποθέσει για μα: συμφωνία αεροπλοεία και καθεστώ συνδεδεμένου μέλου στο ορίζον Και εκεί μπορεί να, και τότε μπορεί να συνεχιστεί η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Για, το ενδεχόμενο, για την ενδεχόμενη συνεργασία. Εγώ, ξέρετε, εργάζομαι στην ε, Digimove, όπου κοιτάμε όχι εμείς μια άλλη μονάδα για την μετα... μετάβαση στο... και χρήση του σιδηροδρόμου, Έτσι λοιπόν και για τα και στα αεροπλάνα αλλά και στους σιδηροδρόμους μπορούν να έχουν εφαρμογή δύο αυτές κοινέ επιχειρήσεις και μπορούμε και να εξασφαλίσουμε ένα ποσοστό του προϋπολογισμού για αυτή τη μορφή συνεργασίας ή κοινέ ε, πρωτοβουλίες, αλλά εν πάση είναι κάπως πρόωρο το να σας ε, δώσω προβλέψεις για το μέλλον. Πάντως, μέσα από αυτήν την κοινή επιχείρηση επεξεργαζόμαστε και με βάση εκτιμήσεις που έχουμε πρόγραμμα δράσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ε, διαχείριση με βάση αξιολόγηση και δημοσιονομικό έλεγχο για να έχουμε και καλύτερη ε, εποπτεία από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τα όσα ε, πραγματοποιούνται μέσω της κοινή επιχείρησης, γιατί λαμβάνει όλο και μεγαλύτερη σημασία το θέμα αυτό και πρέπει βεβαίως και εμείς που λογοδοτούμε σε εσάς να ξέρουμε να δώσουμε απαντήσεις ε, συγκεκριμένες για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εποπτεύει τις ε, κοινέ επιχειρήσεις. Σύντομη απάντησή μου, αλλά ε, δεν ε, έχω περισσότερο χρόνο. Ο Πρόεδρο, ευχαριστώ. Περιμένω να κατακλειστούμε από εκατοντάδε μέλη τη Επιτροπή του Προπολογισμού, αλλά ίσω η συγγήτρια μπορεί να πει δύο λόγια. Έχει το χρόνο. Κυρία Τλαμπάγιουβα. Με εξάφνησε του γεγονό ότι μόνο Τσέχοι μίλησαν. Να πάει λοιπόν ε, η διαχείριση των κυρών επιχειρήσεων, Τσέχη και η Δημοκρατία, τέτοια υποστήριξη που έχετε. Λοιπόν, για να δούμε την πραγματική, το πραγματικό αντίκτυπο και τη σημασία αυτών των ε, επιχειρήσεων θα πρέπει να περάσει και άλλος χρόνος, να κλείσουν και άλλα προγράμματα. Αλλά θα έχουμε τους κύριους δείκτες ε, επιδόσεων για τις κοινέ επιχειρήσεις και στη διαχείριση ε, και στη διατύπωση της έκθεσης. Αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ για το μέλλον είναι ότι θα προβλέψουν την εξασφάλιση του χρόνου την οποία θα ζητήσω διαπραγματευόμενη από την γραμματεία της Επιτροπής μας. Σας υπόσχομαι λοιπόν ότι την επόμενη φορά θα έχουμε πιο πολύ χρόνο στη θέση μας. Ο Πρόεδρος ευχαριστώ την εισηγήτρια, ευχαριστώ τις κοινέ επιχειρήσεις, το Ελεκτικό Συνέδριο, την Επιτροπή για τη συμμετοχή τους Λυπούμε ιδιαίτερως που δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Λυπούμε που χρειάστηκε να σας πιέσω. Αλλά και με την πίεση που σας άσκησα πάλι ξεπεράσαμε το χρόνο μας κατά 10 λεπτά. Ας το λάβουμε υπόψη αυτό για μελλοντικές συνεδριάσεις. Ευχαριστώ πολύ.